Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα να σας ανακοινώσω τις αποφάσεις των συντονιστών. Τις έχετε λάβει βέβαια. Αν μέχρι τις 3 δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Τώρα, λευκή βίβλος για τις μεταφορές. Βιμ Βαντενκάμπ εισηγητής και επειδή είναι ήδη εδώ θα του δώσω το λόγο να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Κύριε Πρόεδρε σας κατευχαριστώ και σας εύχομαι όλους καλημέρα διότι ή έχει βγει ο ήλιος, ήρθε η άνοιξη και λαϊδούν τα πουλάκια. Σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω το έγγραφο εργασίας της μεσοπρόθεσμης παραναθεώρησης. Ε, Λευκή Βίβλος Μεταφορές 2011. Όσοι το κοιτάξατε θα είδατε ότι μαζί με το προσωπικό επεξεργαστήκαμε ένα συνδυασμό μεταξύ καινοτομίας και συνέχειας. Μπορεί να ακούγονται μεγαλεπίβολα όλα αυτά, αλλά αυτή η Λευκή Βίβλος του 11 είχε όντως εφαρμοστεί και θα μπορούσε απλώς να αντιγράφει όλα εγώ δεν αντιγράφει. Το έγγραφο εργασίας έχει ορισμένα στοιχεία συνέχειας στοιχεία δηλαδή που πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε όπως την βιωσιμότητα και το shift, modal shift για τις συνδυασμένες μεταφορές. Αλλά υπάρχουν και στοιχεία καινοτομίας όπως τα λεγόμενα έξυπνα μεταφορικά μέσα, πιο γρήγορες διασυνδέσεις με το ίντερνετ και Έχω 7 γενικά παρατηρήσει, αυτή ήταν η πρώτη. Δεύτερη. Αποφάσισα να αλλάξω λίγο το υπόδειγμα, το πρότυπο. Καταρχήν η οικονομική που τυχεί. Ο τομέας των μεταφορών είναι σημαντικός για την οικονομία μας και πολλοί, πολλοί θέλουν να ασχοληθούν με αυτόν επαγγελματικά. Με ένα λογικό εισόδημα. Γι' αυτό και εγώ τόνισα αυτό το οικονομικό. Τρίτον, κύριε Πρόεδρε μου, ο συνσυνδυασμός ή το λεγόμενο modal shift. Η βάση του Λευκής Βίβλου του 11 ήταν ότι, ό,τι λέγω, Θέλουμε να απομακρυνθούμε από τις αεροπορικές και οδικές μεταφορές για να προωθήσουμε τις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές διάφτες. Μέχρι σήμερα όμως αυτή η μετατόπιση δεν έχει γίνει, δεν έχει επιτευχθεί. Ας πούμε, οι θαλάσσιες μεταφορές ή ποτάμιες μεταφορές δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Θα ήθελα λοιπόν στο έγγραφό μου να τονίσω ιδιαίτερα τον συνσυνδυασμό μάλλον παρά το modal shift. Κύριε Πρόεδρε, τέταρτη παρατήρηση. Αυτό θέλω να το κάνω μέσω της προώθησης ορισμένων πραγμάτων και όχι με ζημίες που θα προκαλούσαμε ή κυρώσεις ή τιμωρίες ή υψηλότερα ποσά και κόστη αλλά μέσω μέτρων που να προωθούν, να δίνουν κίνητρα. Έπειτα η καινοτομία κύριε Πρόεδρε μου είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις μεταφορές. Πολύ σημαντικό. Στο έγγραφο εργασία ε, βάλαμε τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν και την καινοτομία. καινοτομία. Γιατί εγώ βλέπω μεγάλη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και διοδίων. Βέβαια δεν χρειάζεται εδώ να αρχίσουμε ξανά από την αρχή ολόκληρη συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά να δούμε τι επικουρικότητες μπορεί να εφαρμοστούν και γι' αυτό και πώς θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά χάρη στην καινοτομία. Έκτη παρατήρηση προτελευταία για τις κλασικές υποδομές. Βλέπουμε ότι μετά από το modal shift πέρα από το modal shift, οι κλασικές υποδομές δηλαδή οι σιδηρόδρομοι ας πούμε και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές χρειάζονται καινοτομία και ανανέωση των υποδομών τους. Δεν γίνονται όλα από τα ταχύτατα φορτηγά και τα αεροπλάνα, αλλά υπάρχουν και οι κλασικές υποδομές και πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτές και με την κατάστασή των διότι πρέπει να υπάρξει μια συντήρηση σε μερικές χώρες η κατάστασή τους είναι επικίνδυνη όπως στη Γερμανία και πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη μας. Μετά, τελευταία παρατήρηση, η συντήρηση των υποδομών, των κλασικών υποδομών συνδέονται και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ. Και έχουμε ορισμένους φόβους και ανησυχίες ως προς τα κονδύλια του και το πώς θα χρηματοδοτηθεί. Να δούμε λοιπόν αν και με αυτήν τη λευκή βίβλο μπορούμε τίποτε να παρατηρήσουμε. Τέλος δε η βιωσιμότητα γιατί ξέρω ότι είναι από τις έννοιες που σας αρέσουν ιδιαίτερα Πρέπει λοιπόν να είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πολύ το τελευταίο σας σχόλιο για τη βιωσιμότητα, γιατί συμφωνούμε από αυτού. Και σίγουρα πρέπει να είναι προτεραιότητα στο σύστημα. Ο Κλάουντιο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το πολύ καλό του κείμενο. Πράγματι, το μέρο των μεταφορών είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Έχει πολλέ διαφορετικέ παραμέτρου και διαστάσει. Και ευτυχώ οι προτεραιότητέ μα αντικατοπτρίζονται στο κείμενο του κυρίου Φάντεγκαμπ. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Την ίδια στιγμή με την αναθεώρηση τη Λευκή Βίβλου για τι μεταφορέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Λευκή Βίβλου το 2011. Η διαδικασία αυτή που ξεκίνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγε μέρε, με τι διαβουλεύσει με του ενδιαφερομένου, ε, είναι σημαντική. Και βαδίζει παράλληλα με την έκθεσή μα που ελπίζουμε να συνεισφέρει στην πανευρωπαϊκή αυτή θεώρηση τη Λευκή Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο για την πολιτική των μεταφορών, η συγκυρία είναι καθοριστική. Βρισκόμαστε σε ένα τεσταυροδρόμι και η ιδέα της υλοποίηση αλλά και τη κλώση των στόχων τη Λευκή Βιβλίου είναι κάτι που να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Θέλουμε λοιπόν λειτουργική, ευφυή και αποδοτική προ τη χρηστών πόρων ε, πολιτική μεταφορών που θα αναζωογονήσει την οικονομία την οικονομία που έχει πληγεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τη λιτότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ στην προσέγγιση μα και το έγγραφο που προτείνεται σήμερα πρέπει να υλοποιηθεί σύντομα και γοργά όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Ω εισηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχω κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει για τι προτεραιότητε τη ομάδα μου. Θα τι ε, χωρίσω σε τρει κατηγορίε. Πρώτα απ' όλα κοινωνική διάσταση. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή που έχει προβλέψει την κοινωνική διάσταση, η οποία είναι προτεραιότητα για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε το θέμα της εναρμόνισης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις μεταφορές είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την πιστοποίηση και για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις μεταφορές. Ε, στην επικράτεια, ε, στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση. Επίσης δεσμεύομαι να παρακολουθήσω και να προτείνω προτάσεις που θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες ε, αναφορές για την έκθεση. Ως προς τις υποδομές θέλουμε αποτελεσματικές και ευθύες υποδομές. Δεν είναι μόνο απαραίτητες επενδύσεις στις υποδομές, ε, αλλά μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις για μια σειρά από γενιές, για ένα μακρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας και κέρδος, αλλά και η μόχλευση, η, του τέσσερα, του, τετραπλή μόχλευση στο ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα κατάλληλα δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται επαγγελματικά. Επίση έχουμε ένα θέμα με την αιωλική ενέργεια. Χρησιμοποιούμε δημόσιου πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές και πρέπει να έχουμε μια ορθή προσέγγιση. Πρέπει να δούμε λοιπόν Πρέπει να αναζητήσουμε τον σωστό τρόπο να αξιοποιήσουμε τις υποδομές, να είναι μια... να βρούμε μια ε, προσέγγιση που να επιτρέπει να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Αμοιβαίως υποφελεί. Πρέπει να έχουμε έναν ορθολογικό, ορθολογιστικό τρόπο προσέγγισης για την βιωσιμότητα και την απαλλαγή από τον άνθρακα. Ε, Πρέπει να δούμε ως ευκαιρία την ε, ανανέωση του συστήματος μεταφορών και να υπάρξει μια προτεραιότητα σε όλα τα δίκτυα των μεταφορών. Βεβαίως, θα επικεντρωθούμε και στην προστασία του περιβάλλοντος, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάποια στοιχεία ούτω ή άλλω υποφελούνται από τη στήριξη των ιδιωτικών ταμείων, αλλά η μεταφορά πρέπει να αξιοποιείται σε όλε τι παραμέτρου των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε όλου του τρόπου μεταφορά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έτσι θα υπάρχει αυτή η πολλαπλασιαστική επίπτωση και η στήριξη τη οικονομία για την απαλλαγή από τον άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντο. Τελευταία διάσταση που θέλω να το τονίσω είναι η συνολική προσέγγιση αυτή τη έκθεση. Διότι εάν επικεντρωθούμε μόνο στον τομέα των μεταφορών, ξεχνάμε ότι οι μεταφορέ συνδέονται άμεσα με την οικονομία και την ενέργεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική, ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών από την άποψη τη χρήση των πόρων και μια στενή διασύνδεση τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενεργειακή Ένωση και τη στρατηγική μα για, για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Μεταφορών Θα πρέπει επίσης να δούμε την κινητικότητα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να εξυπηρετηθούν επιτέλους και οι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα των μεταφορών να το δούμε ως ένα σύστημα πολυεπίπεδο, ε, συνολικό. Θα πρέπει εμείς να παρέχουμε πολλαπλές υπηρεσίες στους χρήστες και εκείνοι να διαλέγουν το μέσο μεταφοράς που είναι για αυτούς το πιο κατάλληλο. Επίσης θα πρέπει να επιδιώξουμε κάποια συμβιβαστική λύση για τα είδη κινητικότητας που θα προάγουμε και να δώσουμε έμφαση στην αστική κινητικότητα. Διότι εδώ προξενούνται τα περισσότερα προβλήματα, κυκλοφορικά, ε, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η κίνηση στις πόλεις, η χρήση των θέσεων στάθμευσης, και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, κάτι που επίση αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή μα και για μένα προσωπικά, να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει οδική ασφάλεια στι μεταφορέ και κυκλοφορική ασφάλεια. Πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν και με τα θέματα τη οδική κυκλοφορία. Να ε, ευχηθώ καλή επιτυχία στου συναδέλφου που συντάσσουν αυτή την έκθεση και περιμένουμε τι συνεισφορέ και τι προτάσει αλλά και τι των υπόλοιπων συναδέλφων γιατί θα θέλουμε το έγγραφο αυτό να είναι πραγματικά χρήσιμο και να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα έγγραφο που συνδέεται στενά με την αναθεώρηση της Λευκής Βιβλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου καλέσαμε την Επιτροπή να υποβάλει νέε νομοθετικέ προτάσει για σωστή και αποτελεσματική υποτίληση, ε, υλοποίηση του συστήματο μεταφορών που θα αφαιρέσει του πάντε. Ευχαριστούμε τον Μάσο Πορέμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την τιμή σήμερα να μιλάω ξενόματος του Λοτόφσκη και εγώ του συζητητή της ομάδας μου και θα σας παρουσιάσω τις δικές του απόψεις. Καταρχάς θέλω να πω ότι η αναθεώρηση της, επιλογή, της εφαρμογής της Λευκής Βίβλου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δούμε την ευρύτερη εικόνα, ποιος είναι ο στόχος του εγγράφου αυτού. Χαίρομαι γιατί ο εισηγητής έχει λάβει διάφορες απόψεις ε, υπόψη, αλλά έχουμε και κάποιες ε, κριτικές σε ό,τι αφορά τη μείωση του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την κατάρριση της χρήσης παραδοσιακών καυσίμων από τον τομέα των μεταφορών, όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί. Το αντίθετο μάλιστα, όσο δεν τον εξυγχρονισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες, μπορεί να οδηγήσει σε κρίση στον τομέα αυτό. ή δεν γίνεται με σωστό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ποια είναι τα αναλλακτικά καύσιμα και βλέπουμε ότι σε αυτά, στον κατάλογο τουλάχιστον που βλέπουμε, δεν είναι το σχιστολιθικό αέριο, που θα μπορούσε να είναι όμως φτηνή και φιλοπεριβαλλοντική πηγή ενέργειας. Ένα άλλο θέμα είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τις ιοδρομικές μεταφορές, έχει επιτευχθεί πρόοδος. Ενώ στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχουμε επιδοτήσει σε εταιρείε εκτό Ένωση. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για ελεύθερο ανταγωνισμό. Και στι οδικέ μεταφορέ βλέπουμε όλο και περισσότερα παραδείγματα περιορισμού του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, σε κάποια κράτη-μέλη λαμβάνονται μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι μεταφορές στην Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι λόγω της παραμέλης, αν θέλετε, αυτού το τομέα από τους επενδυτές. Δεν σα άκουσα, λέει ο πρόεδρο. Ε, γιατί κάποιοι μιλάνε εκεί πίσω. Λοιπόν, παρακαλώ, μην τα γαδάκια για να ακούμε τον μιλητή. Ο κύριο Πορέμπα. Ναι, υπάρχει και η πολιτική κατάσταση που βλέπουμε στα ανατολικά σύνορα αυτή την περίοδο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα μεταφορά και τις Υπάρχει στρατηγική σημασία πλέον. Πρέπει να προσέξουμε τις μεταφορές, άρα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό το κείμενο για να δούμε πραγματικά κατά πόσον εφαρμόζεται και επιτυχάνει τους στόχους του. Η ομάδα εργασία με συμμετοχή του και ο συγκεκριτή τη ομάδα μου θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ Γκεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάντεν Κάμπ. Συναντηθήκαμε μεταξύ σκιωδών εισηγητών για να επεξεργαστούμε αυτό το έγγραφο εργασία και ήταν πολύ καλή συνεργασία. Είδαμε ότι πολύ λίγε είναι διαφορέ. Όχι, εντάξει, υπάρχουν, υπάρχουν, δεν ανησυχείτε, υπάρχουν διαφωνίε μεταξύ μα, κύριε Πρόεδρε. Απλά όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό στο μέσο να μεταφορά την αγορά, την εννέα αγορά. Είναι σαφέ αυτό. Και Επίση, για το πρόγραμμα εργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι σημαντικό μέσο των μεταφορών. Τώρα, στέφα την ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση, πολύ σωστά τα είπε και η συγητή. <clears throat> Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία θεωρώ καλά και θα ήθελα να συμπληρώσω και κάποια άλλα. Είπε ο ότι κάθε ε, τρόπος μεταφράσης πρέπει να βελτιστοποιηθεί και συμφωνώ. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ό,τι και αν κάνουμε για τη τροπικότητα συνδυασμένες τα κτλ. Κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός από μόνος του θα αυξηθεί ο όγκος των μεταφορών και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργεί η εσωτερική αγορά και για να μείνει η Ευρώπη σε καλή θέση. Καλό είναι λοιπόν που ο Βιν αναφέρει και τα πολύ μακρά φορτηγά οχήματα σε κάποιους τομείς είναι δυνατόν να έχουμε οικολογική ε, προσέγγιση για να μετατοπιστεί το βάρος των μεταφορών από τις οδικές αρτηρίες. Πρέπει να επανέλθουμε στην έκθεση Λάιχτφριντ και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να έχουμε κοντέινερ 48 ιντσών στις ε, θάλασσες. Πώς θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά τα κοντέινερ αν δεν έχουμε συνδρομική διασύνδεση. Με το modal shift συμφωνώ, πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν είναι και τόσο ρεαλιστική. Να περάσουν ε, ε, όλα από τις πλατές μεταφορές ή τις συνδρομικές μεταφορές αντί των οδικών είναι ένας ε, ξιέπαινος στόχος, δεν είναι εφικτός όμως. Ούτε μπορούμε τόσο γρήγορα να φτιάξουμε παντού ε, ράγες και να εκμεταλλευτούμε όλα τα κανάλια και όλους τους ποταμούς. Και θα πρέπει να δούμε και τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου, άρα δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό να μιλάμε για διατροπικότητα συνδυασμένες μεταφορές. Καλά είναι όλα αυτά, καλά κάνουμε και τα αναφέρουμε για το καμποτάζ και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, εσωτερική ναυσιπλοεία. Τα είπε και ο εισηγητής μας. Ήρθε και ο Πίτερ Βαντάλεν που είναι υπέρ των ε, ποταμίσιων μεταφορών. Καλό είναι γιατί μιλάμε πολύ για τις συνδρομικές μεταφορές και όχι για τις πιλωτές. Κάποιες χώρες σίγουρα δεν έχουν ε, δυνατότητες ιστορικής ναυσιπλοΐας, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα model shift. Νέες τεχνολογίες και αυτό είναι σημαντικό. Όταν κάνουμε μια αναθεώρηση να βλέπουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση, τι καινοτομίες υπάρχουν πού και πώς μπορούμε να τις αναφέρουμε. Ο εισηγητής μιλάει για το λεγόμενο tube transport. και τη δυνατότητα χρήσης τελεφερίκ. Πρέπει να υπάρξει επίσης ε, μια αναθεώρηση και των κανονισμών για τα διευρωπαϊκά δίκαια στον τομέα των μεταφορών και για το Connecting Europe Facility. Και έχουμε και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων που το συζητάμε και συζητάμε στο πλαίσιο αυτό και αυτά τα δύο που προανέφερα, τα ευρωπαϊκά δίκτυα Connecting Europe Facility. Πρέπει να ακολουθήσουμε οικολογική προσέγγιση, θα τα συζητήσουμε και πάλι. Είχαμε κάνει και χθε μια πρώτη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και έχουμε και την αρχή ο Ριπένον πληρώνει. Θα μπορούσαμε ίσως τη Λευκή Βίβλο να Μιλάμε και για ένα εναρμονισμένο σύστημα διοδίων για να μπορούμε να έχουμε έσοδα φορολογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ. Για τις, τους συνεργασία αναφέρθηκαν και άλλοι. Εγώ είμαι σκιώδης εκ μέρους της Γκουε και γι' αυτό θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει και όλοι είμαστε πρόθυμοι <clears throat> να εξυγχρονιστούμε ιδιαίτερα για τα κλιματολογικά και την ψηφιοποίηση. Πρώτα για την μείωση των εκπομπών στις μεταφορές. Αυτό δεν μπορεί να περιμένει. Οι κλιματολογικές αλλαγές ε, δημιουργούν προκλήσεις για όλο τον τομέα των μεταφορών. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να περικοπούν εκπομπέ και για τη μεταφορά εμπορευμάτων και για τη μεταφορά επιβατών. Διότι είναι γνωστά, γνωστό ότι είναι, βλάπτουν πιο πολύ εκπομπές διοξιδίου από ότι ακόμη και τα ατυχήματα τα οδικά. Και άρα πρέπει να γίνει κάτι ήδη από τώρα για πρασινότερες μορφές ενέργειας. Η Λευκή Βίβλος του 11 ήδη έθετε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκαπομπών Δυστυχώς ήταν λόγια και όχι πράξεις και πρέπει να κάνουμε μια νέα αξιολόγηση της εργαλειοθήκης μας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεύτερον, η ζήτηση θα έχει επί της θα υπάρξουν επιπτώσεις ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερες ανάγκες μετακίνησης ανθρώπων. Υπάρχει αυτοματοποίηση των εχθρών και τα λοιπά. Η ψηφιοποίηση δεν είναι ο εχθρός μας αλλά φίλος μας. Και με το θοπευτικό του χέρι μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε τα προβλήματα της αποδοτικότητας των μεταφορών η ιδέα αυτοματοποίηση αναμένεται να κάνει τις μεταφορές ασφαλέστερες. Υπάρχουν και νέες μορφές ε, μετακινήσεων όπως το μοίρασμα αυτοκινήτων κλπ. Με λιγότερες συμφορήσεις και λιγότερες εκπομπές. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα δεδομένα που αφορούν με βάση μάλλον τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Δημιουργούνται και νέο τύπου επιχειρήσεις με την ψηφιοποίηση και στις μεταφορές. Και άρα μόνο ένα θέμα συζητιέται πια. All new transport services. Το Uber, Uber διότι πάρα πολλοί θέλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν το σύστημα των μεταφορών στην Ένωση πιο αποτελεσματικό και να αυξηθούν έτσι και οι θέσεις εργασίας ή απασχόλησης. Δυστυχώς οι παραδοσιακοί παράγοντες στην αγορά αυτή αντιδρούν αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι και στην Ευρώπη μόνο υπάρχουν ήδη 15 με 20 εκατομμύρια που χρησιμοποιούν κάποιο είδους ε, μοίρασμα αυτοκινήτων άρα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ζήτηση για αυτόν τον τρόπο μετακίνησης που δεν ικανοποιείται από τους παραδοσιακούς παράγοντες Πρέπει λοιπόν και οι νομοθέτες να δουν αν θέλουν να προστατέψουν μόνο την υπάρχουσα παραδοσιακή δομή της αγοράς των μεταφορών ή αν θα δεχτούν να δώσουν κάποιο χώρο και για αυτούς τους νέους τρόπους μετακίνησης. Εγώ είμαι υπέρ, υπέρ των νέων τρόπων. Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα δουλεύουν όλα αυτά με τον ευρωπαϊκό τρόπο, δηλαδή με πολύ υψηλά πρότυπα ασφαλείας και δίκαιο ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμός στις νέες αυτές υπηρεσίες και αυτό είναι αρνητικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έπειτα ο τομέας των μεταφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν πηγή απάτης για την Ευρώπη. Αν και λένε συνέχεια ότι οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς, αλλά τα ξεχνάμε όλα αυτά όταν μιλάμε για τις νέες ευκαιρίες επιχείρησης, επιχειρήν. Και η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει ο παράγοντας που καθορίζει τα νέα πρότυπα παγκοσμίως τι χρειάζεται να γίνει είναι να παραδεχτούμε αυτά που σας είπα προηγουμένως ότι οι νέοι αυτοί οι τρόποι υπάρχουν να υπάρξει λοιπόν ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις μεταφορές. Δεν θα ήθελα η Ευρώπη να χάσει αυτή την ανταγωνιστικότητα έναντι ασιατικών χωρών ή των ΙΠΑ και τώρα ακριβώς πρέπει να δοθεί αυτή η νέα ορμή. Γιατί αλλιώς θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι μας να τα δούμε ανοιχτό μυαλά και να γίνουν, να εφαρμοστούν και πειραματικά προγράμματα ή όπως τα λέμε εμείς πιλωτικά. Ευχαριστούμε Μπάσε Εκάουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βιμ Κάμπ για αυτό το πρώτο έγγραφο συζήτηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Βαντεν Κάπ ε, που μας παρουσίασε τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε αυτό το έγγραφο, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο τι κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Θέτει κάποια στήματα επιτάκτως, αλλά βέβαια τελικά πρέπει να βρούμε μια κατεύθυνση. Αλλιώς θα μείνουμε σε ένα συμβιβαστικό έγγραφο άτομο και θα πάμε στην επόμενη έκθεση. Εγώ δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Αρκετά έγγραφα έχουμε συντάξει για το μέλλον τα Και, και θα μπορούσε και η Επιτροπή να συντάξει πολλές ακόμη λευκές βίβλες για τις μεταφορές. Το θέμα είναι να αλλάξει κάτι. Άκουσα προσεκτικά λοιπόν τον κύριο Βαντενκάμπ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι είπε για τη βιωσιμότητα, όπως το διατύπωσε. Είπε ότι εστιάζω λίγο περισσότερο στην οικονομία και λίγο λιγότερο στη βιωσιμότητα γιατί χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας. Είναι ένα παλαιού παραδείγματος ε, στο οποίο βρίσκεται ακόμη ο κ. Βαντενκάμπ. Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες αναλεκτικές. Και επίσης η βιωσιμότητα λέτε πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ε, λέτε το αυτονόητο και συμφωνώ και εγώ. Ε, Αυτό λέμε κι εμείς. Είναι σημαντικό η βιωσιμότητα και αν δεν αλλάξει δεν θα έχουμε μέλλον στις μεταφορές. Δεν τα κατάλαβα πολύ καλά αυτά τα σχόλια. Ας γίνει λοιπόν κομβικό θέμα το θέμα της βιωσιμότητας. Και βέβαια θέσεις εργασίας πολύ επιθυμούμε. Είναι ένας άλλος στόχος. Θέλω να πω και κάτι ακόμη μια επισκόπηση για το που είμαστε με αυτή τη λευκή βίβλα. Αν αυτός είναι ο στόχος, νομίζω ότι ε, πρέπει να δώσουμε μια αίσθηση κατεπίγοντος. Από την ανακοίνωση και μετά προέκυψε μια τεράστια κρίση. Το να προσποιούμαστε, ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, στο 2007, ήταν πολύ ωραίος ο κόσμος μας πριν την κρίση, αυτό δεν λειτουργεί. Απ' την άλλη, αν δούμε τις προκλήσεις, παραδείγματος χάρη, αλλαγή του κλίματος, αυξάνονται οι μεταφορές. Είναι ο μόνος τομέας που αυξάνεται. Γι' αυτό πρέπει κάτι να αλλάξει. Μέχρι τώρα, αν δεν κανείς τι έχουμε κάνει με όλα αυτά, ε, τα, με όλες αυτές τις δράσεις και με όλες αυτές τις προτεραιότητες, δεν κάναμε και πολλά, δεν έχουν αλλάξει και τόσα. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεργαστεί αυτή την αναθεώρηση, θα μας παρουσιάσει ίσως του χρόνου ένα εντυπωσιακό κατάλογο των αλλαγών, αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Ξεκολουθούν να έχουν πολλά προβλήματα στον τομέα των μεταφορών. Μην κοροδευόμαστε λοιπόν. Ως Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να τα πούμε πιο ξεκάθαρα εμείς τα πράγματα γιατί υπάρχουν και ευκαιρίες. Γι' αυτό και λέω ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική πλευρά μπορούν να συμβαδίσουν. Ψηφιοποίηση, καινοτομία, στο logistics, ε, χρήση αυτοκίνητο περισσότερους ε, του ενός <clears throat> και τα λοιπά. Μην αναζητούμε μόνο παραδοσιακές λύσεις, δεν βοηθά αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και να είμαστε και πιο ε, ε, ρητοί στην ε, διατύπωσή μας. Ούτε και στο model shift λοιπόν και πολλά. Είπε και ο Βαντενκάμπ θέλει περισσότερη ανταμοιβή και λιγότερη τιμωρία. Ερώτηση προς τον εισηγητή. Τι εννοείται ακριβώς. Αυτή τη ανταμοιβή δεν ξέρω πώς να αντιλαμβάνεις ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται ακριβώ. Ελπίζω η τιμωρία, όπως την λέτε, να μην είναι απλά το να τακτοποιήσουμε τα θέματα της τιμολόγησης με τις διάφορες, με τις διάφορες τρόπους μεταφοράς. Εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει ισομέρης κατανόμη. Αν δεν γίνει σωστά, τότε θα παραμείνει και το modal shift θεωρία και δεν θα περάσουμε ποτέ στην πράξη. Το πρόβλημα της τιμολόγησης είναι τεράστιο. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο επικρίτικοι στον τομέα αυτό. Δεν είναι μόνο για άποψη των πρασίνων. Αν πιστεύεις την αγορά όπως πιστεύεις, Βιν, θα πρέπει να συμφωνήσει μαζί μου ότι πρέπει να πάει και σωστή τιμολόγηση και ομοιομορφία στις τιμές. Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτή τη λευκή βίβλο με την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μια τεράστια πρόκληση. Έχουμε έκθεση λοιπόν για το θέμα αυτό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μπορούμε να συσχετίσουμε τα δύο θέματα πιστεύω και πρέπει να το κάνουμε. Κοινωνική διάσταση. Χαίρομαι ιδιαίτερος που το πρόσθεσε αυτό το θέμα ο εισηγητής. Τι όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση για μια συμπεριφοριστική αλλαγή αν θέλετε. Αν λάβουμε υπόψη μας σοβαρούς αυτές τις αλλαγές δεν μπορούμε απλά να προτείνουμε τις τεχνικές λύσεις, νομίζω ότι θα τα λύσουν όλα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση περί συμπεριφοριστικής αλλαγής. Και στην Κομισιόν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν λέω ότι θα αλλάξει αύριο η Ευρώπη με αυτό. Αλλά αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Ούτε εθελοτυφλώντας μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και στο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε αρχικά τον κύριο Φάντερ Κάμπ. Είναι πολύ καλό το σχέδιο έκθεση του, έχει θέσει τι σωστέ προτεραιότητε και έχει κάνει μια πολύ σωστή ανάλυση του θέματο. Εδώ έχουμε όμω μια σειρά από στόχου για το 2050. Βεβαίω απέχει αυτή η ημερομηνία, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τι σωστέ προτεραιότητε. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία. Έχουμε πλέον ε, πολλά κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Η ενιαία αγορά προκαλεί προβλήματα σε εθνικό επίπεδο ως προς το κοινωνικό ντάμπινγκ και βλέπετε πως η Γερμανία προσπαθεί να προβλέψει τον κατώτατο μισθό. Αυτά είναι φοβερές αλλαγές. Για τη βιωσιμότητα. Βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα των δίκαιων κανόνων. Διότι τον ανταγωνισμό κάποιε φορέ τον ε, εκμεταλλεύονται εργοδότε για να επιβάλλουν πολύ, πολύ κακές συνθήκες. Έτσι λοιπόν οι εταιρείε υποχρεούνται να έχουν πολύ αυστηρές πολιτικές πρόσληψεις λόγω του στιγνού ανταγωνισμού, ενώ κάποιες άλλες δεν καταφέρνουν καν να αναδυθούν και να λειτουργήσουν στην ενιαία αγορά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις εταιρείες που έχουν τις ε, καλύτερες πολιτικές πρόσληψης και τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, δημιουργώντας την αγορά μας, να μην καταστρέψουμε τις ε, εταιρείες αυτές. Για τις εκπομπές λοιπόν φαίνεται να μην μειώνονται τόσο όσο επιδιώξαμε. Είναι αρκετά σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε ότι όλα αυτά γίνονται για τους πολίτες που συχνά δεν ε, καταφέρνουν να εξυπηρετηθούν. με αυτά που τους προτείνουμε. Υπάρχει και το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα. Αλλά ανησυχώ που θα καταλήξει και που θα μας οδηγήσει. Νομίζω ότι τα θεμέλια του δεν είναι και τόσο αδιάσυστα. Θα πρέπει να σκεφτούμε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των μεταφορών, ε, γιατί πολύ συχνά ακούμε να μας κατηγορούν για τάσεις προστατευτισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Δεν είναι το πρόβλημα εδώ αν υπάρχει προστατευτισμός ή όχι. Μα ενδιαφέρει οι πολίτε μα να μπορούν να έχουν μια ε, εύκολη διαβίωση σε αυτέ τι συνθήκε. Δεν θέλουμε να τους δεσκεράνουμε με τον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει και την ενέργεια να τη θέσουμε στην υπηρεσία της αντιμετώπισης αυτού του είδους των φαινομένων. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, πρόβλεψης νέων κανόνων ξανά και ξανά. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχοντες κανόνες τουλάχιστον ε, υλοποιούνται. Και να θυμόμαστε ότι υπάρχουν καθημερινά πολίτες που υπάρχουν θύματα εκμετάλλευσης από στιγνού εργοδότες. Πρέπει να επιφερθούν βελτιώσεις και να επιβάλλονται σωστά οι κανόνες σε μια αγορά που θέλουμε να είναι δίκαιη. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή μας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Όσα προβλέψαμε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες ε, μπορούν να μετακινούνται ε, με ένα τρόπο που να μην είναι ακριβώς, υπερβολικά ακριβώς. Πώς να αξιοποιήσουν ε, τα μέσα μεταφοράς που τους προτείνουμε πολίτες αν δεν μπορεί να τα πληρώσει τσέπη του. Έτσι λοιπόν, όπω είπε αυτή εξ αρχή, το έγγραφο του κ. Βαντονκάμπ είναι πολύ καλή βάση εργασία για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν του κοιόδη εισηγητέ και έχουμε και άλλους 8 στον κατάλογο. Και ο Σμάιλερ του 8 λεπτά, τέρμα. Α, και ο Φαντάλεν. Κλείνω κατάλογος όμως τώρα. Τζάκι Φώστερ, 3 λεπτά. Είστε η πρώτη κυρία Φώστερ. Yes, of course. Δεν σας ξεχνάω ποτέ. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, νόμιζα ότι θα πάρετε τις ομάδες με τη σειρά. Ναι, νόμιζα θα περάσετε από το ΕΛΚ στους σοσιαλιστές και... Στο δεύτερο γύρο είναι ελεύθερα τα πράγματα. Είσαστε πρώτοι. Νομίζω ότι πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ακούσαμε. Πρέπει να πούμε αρχικά ευχαριστώ προς τον εισηγητή γιατί είναι πραγματικά ευρύτατη η έκθεση του, αλλά αυτό που δεν βλέπω και επειδή το παλιότερα μέλη αυτή τη Επιτροπή, από το 99 συγκεκριμένα, βλέπω να γίνονται πολλά σχόλια από συναδέλφους εδώ και δεν έχουμε κάνει τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια ως προς το πώς θα βελτιώσουμε τις μεταφορές και πώς θα προωθήσουμε και άλλα θέματα ταυτόχρονα. Πρέπει να προσέξουμε όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής ε, τη, τα τελευταία 15 χρόνια να μην λέμε ότι δεν έχουν κάνει και τίποτα, δεν καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχουν ε, γίνει πολύ καλές νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες για τις εισοδικές μεταφορές, για τους σιδηροδρόμους, Μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε αποφάσει και για τα επόμενα 15 χρόνια, αλλά αν δούμε τι γίνεται με τι πρώτε μεταφορέ, την αεροπλοεία, του εκδρόμους, έχουμε τεράστια νομοθετήματα που έχουν ε, προβλεφθεί εντωμεταξύ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε είναι η νομοθεσία που ήδη ισχύει να υλοποιείται. Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το συμφωνήσουμε και δεν βρίσκω ε, σκόπιμο όταν κάτι δεν υλοποιείται ορθώς, να διαλέγουμε ένα διαφορετικό δρόμο και να προσπαθούμε να προβλέψουμε ένα άλλο νομοθέτημα για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σε μικροσκοπικό επίπεδο τους πάντες. Υπάρχουν 28 κρατη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ε, τι τις παραδοσιακές τους συνήθειες, τα συστήματά τους που μπορεί να μην είναι τα ίδια με του γείτονα στην διπλανή χώρα. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε τους στόχους της κοινής αγοράς, αλλά δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν έχει κανείς ε, την τέλεια συνταγή για να αλλάξει οι δομές που ισχύουν εδώ και δεκαετίες στα περισσότερα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι κάποιες φορές πολιτική βούληση υπήρξε με σωστές πρωτοβουλίες για τη διασυνοριακή διασύνδεση. Αλλά σε κάποιες ε, περιπτώσεις δεν υπήρξε αυτή η βούληση και δεν έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Επί τη ουσία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Ευθύνε, για να ε, προβλέψουν τις κατάλληλες υποδομές, τους κατάτος μισθού, της χώρε τους, να βεβαιωθούν ότι όσοι εργάζονται στον τομέα μεταφορών ε, εργάζονται με καλές εργασιακές συνθήκες και νομίζω όλα τα κράτη-μέλη ε, αναγνωρίζουν τι συνδικαλιστικέ οργανώσει και ορθώ. Υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει για τις διάφορες εταιρείες μεταφορών, οπότε για τις εταιρείες που δεν ε, ε, έχουν καλές εργασιακές συνθήκες θα πρέπει οι συνδικαλιστές να λάβουν ε, την πρωτοβουλία και να τους προσάγουν στις υπεύθυνες εθνικές αρχές. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να κλείσει αυτό το θέμα και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι καθόμαστε εδώ με τέσσερα χρόνια μπροστά στη θητεία μας και κοιτάζουμε πώς τα έχουμε πάει. Ε, κάποια πράγματα ήδη έχουν αρχίσει να ισχύουν και τα πάμε αρκετά καλά, αλλά ε, αν υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας και θέλουμε να προχωρήσουμε, να σκεφτούμε το Single Sky, τον ενίο ουρανό. Ε, είναι γελία η κατάσταση που έχει προκύψει. Έχουμε 29 κρατημέλη που προσπαθούν να πιέσουν με επενδύσεις που ξεκινάνε από το πρόγραμμα Γαλιλαίο να οδηγήσουν στην αποδοτική λειτουργία του κλάδου. Αυτό το κόστος το πληρώνει ο καταναλωτής και πρέπει το δικό του ανταγωνισμό να τον ε, πληρώσει, να πληρώσει τα σπασμένα. Μπορούμε λοιπόν με περισσότερες πολιτικές κινήσεις να λύσουμε περισσότερα ζητήματα. Να ευχαριστήσω εδώ τον εισηγητή που έθεσε αυτά τα θέματα και να πω ότι πιστεύω θα έχουμε μια λογική συζήτηση. Τζάκι, πρέπει να σε διακόψω, όχι, όχι, έχεις ε, ε, πάει στα δύο λεπτά, δεν έχεις περισσότερο χρόνο. Ο Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι γνωστές οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Πρέπει να κάνουμε την απογραφή μας και πιστεύω πως ο συνάδελφος Εβήμ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική δουλειά, την οποία θα βελτιώσουμε κιόλας. Όπως είπα, είναι γνωστές οι προκλήσεις και πιστεύω πως ήδη έχουν υποθεί πολλά. Η έλλειψη ικανοτήτων, η έλλειψη υποδομών είναι ένα θέμα που παραμένει στο προσκήνιο και αυτή η προσπάθεια να έχουμε λιγότερο άνθρακα είναι μια προσπάθεια που συνεχίζει να υφίσταται και θα μας απασχολεί μέχρι να βρούμε κάποιες ε, σωστές και ξεκάθαρες λύσεις. Για παράδειγμα, η Τζούλη Φώστερ αναφέρθηκε για την αεροπλοεία, όπου έχουμε παραμείνει στάσιμοι και στο μεταξύ οι Κινέζοι φτιάχνουν νέες ε, γραμμές, καθώς επίσης και στις ε, σιδηροδρομικές ε, μεταφορές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας όλες αυτές τις προκλήσεις που θα επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και να προσαρμοστούμε Επίσης, οι κοινωνικές απόψεις, ε, κατώτατος ε, μισθός στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε την νομοθεσία, ωστόσο έχουμε έλλειψη εφαρμογής αυτής της ε, νομοθεσίας και πιστεύω πως ε, θα διαρκέσει πάρα πολύ μέχρι πραγματικά να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Επίσης, συστήματα ασφαλείας των μεταφορών, συστήματα ε, βοήθειας, δεν υπάρχουν όρια στην τεχνολογία, ωστόσο υπάρχουν όρια στην πολιτική βούληση και με δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα των επιβατών, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά, ο κατασκευαστής, ε, η Google, ποιος τέλος πάντων θα τα διαχειρίζεται. Και πιστεύω πως πραγματικά όποιος ξέρει τις προκλήσεις του τομέα, όποιος ξέρει τι χρειάζεται να γίνει και τι λείπει, εκνευρίζεται με αυτήν την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα και άλλους λόγους, όμως όπως είπα έχουν ήδη αναφερθεί από τους προηγούμενους συναδέλφους. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω λέγοντας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ στον συνάδελφο Βιν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μοντέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φάντεν Κάμπ για την σύνταξη αυτού του εξαιρετικού έγγραφου εργασία και για τι πολύ καλέ προτάσει που έκανε. Εδώ να πω ότι σήμερα ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν ενιαίο χώρο μεταφορών στην Ευρώπη, όμως Πώ το 2050, ε, ακόμη και αν δεν το έχουμε καταφέρει, πιστεύω ότι θα έχουμε ανοίξει το σωστό δρόμο. Και θα είναι ένα δρόμο ε, βιώσιμο και με στόχο τη βιωσιμότητα. Ελπίζοντας ότι αυτοί που θα ωφεληθούν είναι αυτοί που είναι και στον πυρήνα τη συζήτησή μας, δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να κάνω κάποια σχόλια που μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά και που ήθελα να αντικατοπτρίζονται στην πρόταση αυτή για την αναθεώρηση της Λευκής Ε, η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τις θαλάσσιες μεταφορές. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρω και την ενίσχυση της δυνατότητας της ανταγωνιστικότητας μάλλον των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους ε, θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους του θαλάσσιου δρόμου, δηλαδή και, και να έχουμε μια ενιαία θαλάσσια πολιτική. Θα πρέπει να την ε, προάγουμε την ε, έννοια αυτή, την όλη αντίληψη και να προτείνουμε συγκεκριμένε δράσεις για να δώσουμε δυνατότητε στην ενιαία θαλάσσια πολιτική. Διότι προ στιγμή νομίζω δεν έχουμε αναπτύξει το δυναμικό που διαθέτουν οι Στο ίδιο πλαίσιο θεωρώ σημαντικό να δούμε πώς έχουν τα πράγματα με τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και στα ευρωπαϊκά λιμάνια και στα σκάφη. Επίσης καλό θα ήταν να πούμε ότι χρειάζεται και κάποια στρατηγική δράση για την διασύνδεση μεταξύ των νήσων. Χρειάζεται μια διορατική στρατηγική που να δώσει σημασία στις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών νήσων της Ευρώπης. Και αυτό με συγκεκριμένες δράσεις. Διότι εδώ έχουμε και συγκεκριμένες περιοχές με πολλούς περιορισμούς στο επίπεδο των μεταφορών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, επειδή είναι εξόχως απόκεντρες, αλλά και το θέμα των νέων τρόπων εμπορίας της μετακίνησης των επιβατών όπως προκύπτουν. Εδώ συζητήθηκε το τι είδους το τι είδου νομοθεσία θέλουμε να προβλέψουμε για αυτού του νέου τρόπου εμπορία των μέσων μεταφορά. Και επίση ένα τελευταίο σχόλιο για τα κοινωνικά και μισθολογικά των εργαζομένων στου σιδηροδρόμου. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αναθεώρηση για αυτά τα θέματα για να αποφύγουμε εξέλιξει όπω οι πρόσφατε και ε, οι απομακρυσμένε περιφερειακέ χώρε, όπω η Πορτογαλία να μην έχουν την ίδια πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει να ξεπεραστούν φραγμοί και διακριτικέ μεταχειρήσει. Και για να ολοκληρώσω να πω ότι όντω ελπίζω να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που τώρα έχουν υποβληθεί και ε, αφού συζητηθούν να έχουμε ένα νομοθετικό έγγραφο που τελικά θα καταφέρει ε, να βελτιώσει αυτό που ακριβώ επιδιώκουμε, τη ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρή Κριστίνα Νοτού. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω πολλά ερωτήματα και πολλές παρατήρησεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση του σε σχέση με τη Λευκή Βίβλου. Καταρχάς, θα συμφωνήσετε μαζί μου κύριε Κράμερ, κύριε Πρόεδρε, ότι ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα δεν αντιμετωπίζεται σωστά ε, Σίγουρα με τις κατάλληλες υποδομές μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές, περιθωριακά όμως. Ε, την μείωση των αχρίαστων μετακινήσεων θα ήταν ο καλύτερος τρόπος. Ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες, δεν είναι ε, μόνο θέματα της δικής μας Επιτροπής Ενθάρρυνσης Τοπικής Παραγωγής, καλύτερη διασύνδεση, προστασία του περιβάλλοντος, περιαστικοποίηση. Επίσης, έχουμε τα θέματα της δυναμικότητας των αερολιμένων. Πολλά αεροδρομία έχω καταθέσει και προφορική ερώτηση, ιδίω επαρχιακά, ε, ξεπερνάνε τις δυνατότητές τους, όπως βλέπουμε στη Γαλλία. Γίνεται υπερεκτίμηση ή πάντων κακή εκτίμηση της κίνησης στα αεροδρόμια. Ε, για τις αεροδρόμους, Πημένουμε στην ανάγκη να ανοίξουμε στον ανταγωνισμό, την αγορά εσωτερικών μεταφορών, ενώ δείχνει η πρόσφατη εμπειρία ότι δεν είναι προσαρμοσμένος ο ανταγωνισμός στη φύση των εσωτερικών μεταφορών και έχουμε πάντα μείωση της ασφάλειας και της ε, ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση τιμής ε, και κατάσταση αρκετά ε, ευάλωτη θα τη χαρακτήριζα για τους διάφορους φορείς. Κυρία Μπιλμπάου, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θα ήθελα όμως στην έκθεση αυτή να περιλαμβάνεται και κριτική και αυτοκριτική και να είναι σαφές αυτό. Η έκθεση αυτή πρέπει πέρα από συγκεκριμένους στόχους, με τους οποίους θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και είμαστε όλοι σύμφωνοι, με κάποιες αποχρώσεις ίσως, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι βιώσιμες, και σίγουρα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους ε, της Λευκής μου, όταν διαβάζω την έκθεση μου λείπει ε, το ερώτημα. Γιατί δεν το πετυχαίνουμε, γιατί δεν πετυχαίνουμε τους στόχους και νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε στα συγκεκριμένα προβλήματα που κάθε μέρα βιώνουμε και στο κοινοβούλιο μας εδώ. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει ακριβώς και μιλώ για την τέταρτη δέσμη μέτρων για τις συνδρομικές μεταφορές που ήταν απαραίτητο γιατί δεν τηρήθηκε το τρίτο πακέτο, θέλουμε ενεργειακή απόδοση, θέλουμε ενιαίους εθέρες. Τα έχουμε γραμμένα όλα αυτά. Σε χαρτί εννοώ. Πρέπει όμως να δώσουμε και ένα σαφές αποφασιστικό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη. Να τους πούμε ότι για να πετύχουν όλους αυτούς τους στόχους χρειάζονται, πρέπει να υιοθετήσει μια διαφορετική διακυβέρνηση των μεταφορών στην Ευρώπη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον να μην τηρούμε συστηματικά αυτά που λένε οι εκθέσεις και να μπλοκάρουμε συνεχώς με αυτή την έννοια εθνικής κυριαρχίας που τον 21ο αιώνα έχει ξεπεραστεί. Πρέπει στην έκθεση αυτή να μιλήσουμε για πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να εκπέψουμε και ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως βέβαια προς το Συμβούλιο. Γιατί Διαρκώ είμαστε αντιμέτωποι με το Σύμβουλο αν θέλουμε να ε, καταρρύψουμε αυτού του φραγμού. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε αν χρησιμοποιούσαμε πιο αποτελεσματικά του πόρου μα. Και έτσι στην Ευρώπη θα δημιουργούσαμε κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο χρειάστηκε να ξαναορίσουμε τα ευρωπαϊκά έργα μεταφορών, ποια είναι τα οι προτεραιότητές μας δηλαδή των μεταφορών και ουσιαστικά εκεί βλέπουμε τα ίδια με το 1994, το Συμβούλιο του ΕΣΥ, του ΕΣΕΝ, της ΕΣΥΣ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία έκθεση και να μην μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα που είναι και το πρόβλημα με επικεφαλαίο. Και μιλήσαμε για την Ιταλική Ασία, τις κοινωνικές επενδύσεις. Πρόσφατα έφτασε ένα σειρμός από την Κίνα στη Μαδρίτη. Αν εμείς ως Ευρωπαίοι δεν μιλήσουμε για την ανάγκη να έχουμε μια άλλη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στις μεταφορές και αν δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να καταλήξουμε αυτούς τους φραγμούς, δεν θα πετύχουμε τους στόχους. Και τέλος, τι θα συμβεί. Θα συμβεί αυτό που άκουσα σε μια ημερίδα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη για τους ενίους εφαίρες, το ενίο ουρανό. Ήρθανε και μου είπαν κάποιοι. Ακούστε, λείπουν πολύ από αυτή την ημερίδα. Γιατί? Εγώ είμαι ένας μηχανικός που 40 χρόνια ακούω να γίνεται λόγος για τον ενία ουρανό χωρίς να έχουμε ακόμη φτιάξει τίποτα. Και γι' αυτό είναι πολλοί κόσμος απογοητευμένος και αυτό δεν ήρθαν σε αυτή την ημερίδα. Πώς επιτεχάνουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους. Ας είμαστε ειλικρινείς και τίμοι. Αν δεν μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα θα έχουμε μια ακόμη έκθεση που θα μοιάζει πάρα πολύ με όλες τις άλλες εκθέσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και όλα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι εργαζόμαστε και είμαστε ικανοποιημένοι και τίποτα παραπάνω. Πρέπει όμως να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα και να δώσουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς το Συμβούλιο και να μιλήσουμε τη γλώσσα της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά του γιατί έχουμε την παρουσίαση της Λευκής που τόσα χρόνια πήρε, τώρα έχουμε αυτή την αξιολόγηση για να κάνουμε με έναν απολογισμό, όπως είπε και η κυρία Μπιλμπάου. θα ήθελα και εγώ να ε, προσεγγίσουμε διαφορετικά κάποια ζητήματα. Σίγουρα είναι δύσκολο να πάρει κανείς απόσταση από πράγματα που μετά που έχει καταπιαστεί έτσι από πολύ κοντά. Εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε το πρόβλημα των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Είχαμε μια μερίδα για την ενέργεια και μας είπαν ότι οι ελεκτές σε πολύ λίγα χρόνια θα εξαφανιστούν και δεν είναι εύκολο να εκπαιδεύσει ε, έναν ελεγκτή, δεν τον αγοράζει στο σούπερ μάρκετ και το ίδιο ισχύει και με τα πληρώματα θαλάμου επιβατών, ε, με τους πιλότους, ε, τους μηχανοδηγούς, των σειρμών, όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε με ένα άνοιγμα αγορέ και όπως και ο κ. Ζαντεκά πρέπει να προσπαθήσουμε το κοινωνικό πακέτο. Τι κάνουμε δηλαδή, με ποιο τρόπο. Το επάγγελμα, τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις μεταφορές θα τα προωθήσουμε λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις επαγγελματικέ διαφορές και να μην το βάλουμε μόνο στο άνοιγμα, αλλά το placing people να το βάλουμε στο επίκεντρο. Δεν θέλουμε μόνο επιβάτες, θέλουμε και εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών. Δεύτερον, ένα άλλο θέμα που μπορούμε να ενισχύσουμε έχει να κάνει και με την ίδια με τις υποδομές και υπάρχουν σημαντικά στοιχεία εδώ που θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Έχουμε προκλήσεις όπως ασφάλεια για τα νέα ε, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά οχήματα, ε, logistics, εφοδιαστική. Πρέπει να υπερπηδήσουμε τα εθνικά εμπόδια. Παραδείγματος χάρη, εγκατάλειψη των συνδυασμένων μεταφορών Σίγουρα λέμε ότι το θέμα είναι να, μειωθεί, να μειωθούν οι ειδικέ μεταφορέ, αλλά δεν αρκεί να το λέμε αυτό. Πρέπει να δούμε και πώ θα γίνει. Υπάρχουν εθνικοί νόμοι που δημιουργούν εμπόδια για την αλλαγή τρόπου μεταφορά, για την κινητικότητα την αστική. Συμφωνώ. Το θέμα των εμπορευματικών μεταφορών, είδα κάποια σχόλια που μου φαίνονται έτσι πολύ φουτουριστικά. αλλά μου σηκώνεται και τρίχα κάγκελο με μερικές ε, προτάσεις. Ασφάλεια. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας οδικών μεταφορών. Υπάρχουν και γενικές απειλές. Έχουμε τα συλλογικά κέντρα μεταφορών, αυτοκίνητα, αερολιμένες και έπειτα. Χρηματοδότηση αναφέρεται μόνο ως charging. Εντάξει, έχουμε τα διόδια και τα άλλα τέλη, αλλά νομίζω ότι εμείς, αυτό που δεν γίνεται και με το πρόγραμμα Juncker, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές και τις μεταφορές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα φτιάξουμε ένα πάζελ. Ένα συνονθήλευμα λύσεων που δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Τέλος, το μοντέλο κινητικότητας. Το είδαμε και στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να σταματήσετε. Ναι, τέλο πάντων έλεγα για αυτό το μοντέλο κινητικότητα. Μάλιστα, πρέπει να σας διακόψω γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν θα μας ε, φτάσει ο χρόνος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Τέλη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την δουλειά του και δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις κριτικές που έχει δεχτεί. Στην τέταρτη σελίδα αναφέρει τους προβληματικούς τομείς. Την απαλλαγή από τον άνθρακα για παράδειγμα. Αναφέρει λοιπόν τα πιο σημαντικά προβλήματα και εκεί όπου χρειάζεται δράση. Επίσης, διαπιστώνεται, και εδώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το έγγραφο, ότι χρειάζεται να γίνει μια τέτοια συζήτηση, όπως και θα γίνει αργότερα σήμερα. Χρειάζεται μια αξιολόγηση των γεγονότων έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους αφιλόδοξους στόχους που αναφέρονται στην Λευκή Βίβλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στόχους μέχρι το 2050. Και μπορεί να μας φαίνεται μακρινή αυτή η ημερομηνία, πρέπει όμως να δράσουμε από τώρα για να προλάβουμε. Χρειάζεται επίσης να δούμε εάν τα συστήματα υποδομών συνάδουν με τις ε, προδιαγραφές της ε, νομοθεσίας και αν συνάδουν με την υφιστάμενη νομοθεσία. Και να δούμε πώς ε, συνδέονται όλα αυτά με τους οικονομικούς δείκτες. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εμβαθύνει με αυτή τη μελέτη και να διευκολύνει έτσι την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. έτσι ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει βασιζόμενη σε αυτά τις μελλοντικές της ενέργειες. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πραγματιστές. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ερτούγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Βάντεκαμπ. Πιστεύω ότι σε αυτές τις 12 σελίδες αναφέρονται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και πραγματικά διάβασα την έκθεση και σημείωσα τα πιο σημαντικά κομμάτια. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή, διότι αρχίζει αναφέροντας τα εναλλακτικά καύσιμα και τις δεσμεύσεις για την εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων για την ποιότητα. Επίσης, θεωρώ εξίσου καλή την αναφορά στην τεχνολογία και στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, διότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν αυτού, η αναφορά στους ε, στόχους των μηδενικών εκπομπών είναι εξίσου σημαντική και θα ήθελα και σε αυτό το σημείο να προσθέσω δύο πράγματα, ότι τα κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερη ευθύνη, διότι αυτά θα κληθούν να εφαρμόσουν και τα μέτρα. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντική την αρχή του οριπένων πληρώνει που αναφέρεται στο κείμενο και αν κατάλαβα καλά ο εισηγητής δηλώνει την επιθυμία του για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από ό,τι λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα προγράμματα και να προωθήσει τις ε, καλές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα καλωσορίσω αυτό το οδικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα η έκθεση αυτή επιδέχεται προσθήκες, για παράδειγμα τις ε, κοινωνικές προϋποθέσεις. Τώρα στη σελίδα 9 βλέπω ότι υπάρχει μία διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και χρειάζονται κάποιες προσθήκες οι οποίες θα δείχνουν τον σαφή προσανατολισμό μας στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης, την αλλαγή μοντέλου. Πιστεύω πως εδώ πρέπει να αναφερθεί η αηφορία και δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε αυτός ο κανόνας των 300 χιλιόμετρων. ο οποίος ε, ήταν ένας κανόνας που έχει τεθεί ήδη από το 2011 και στην σελίδα 11 γίνεται αναφορά στα μακρύτερα και βαρύτερα οχήματα, το οποίο είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα. Εδώ θα ήθελα να προσθεθεί η σαφής αναφορά του ποιος θα επιφορτιστεί αυτή την ευθύνη της αλλαγής. Ο κύριος Βαντάλεν έχει το λόγο. Ε, Δεν μπορούμε να σας ακούμε, παρότι έχετε ανοίξει το μικρόφωνο. Ίσως μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά. Πρόεδρε, θα δοκιμάσω σε αυτό το μικρόφωνο, μάλλον δουλεύει. Πρόεδρε, ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές στον κύριο Φανενκάμπ από τον μεγάλο γερμανό φιλόσοφο, τον Γκέτε. που είπε ότι ο πλέον γνώστης φαίνεται στην τους ε, περιορισμούς και εκεί εξασχεί τη δεξιοσύνη του. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Φαντενκάμπ, ε, στην επεξεργασία, στη σύνταξη της έκθεσης αυτής, περιοριστείτε στα θεμελιώδη και στα βασικότερα, αν θέλετε. Δηλαδή, μην ζητάτε περισσότερους κανόνες, περισσότερες προσαρμογές και περισσότερη νομοθεσία. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εδώ. Ο άδικος ε, και αθέμητο ανταγωνισμός των τομέα μεταφορών. Ιδίως ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές και τις αεροπορικές. Εκεί θα πρέπει να αφοσιωθούμε. Μην ξεκινάτε με ένα κατάλογο νέων ζητημάτων που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και έπειτα, Πρόεδρε, να πω ότι έχουμε πολλούς κανόνες και κανονισμούς σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα στην Ευρώπη έχει να κάνει με την υλοποίηση. Πολλές φορές δεν υπάρχει κατάλληλη υλοποίηση ή η υλοποίηση γίνεται με τρόπο αρκετά αυθαίρετο και μεραλυτικό. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Για τις οδικές μεταφορές λόγου χάρη, δεν μπορούμε να θεωρούμε το δίκτυο στην Ιταλία το ίδιο με τη Γερμανία ή τις κάτω Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικές φορέ μπορεί να χρειάζονται και διαφορετικέ ε, ερμηνείες ώστε να αποφεύγονται οι τρευλωτικές πρακτικές. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες βασικές παρατηρήσεις πρόεδρε που πρέπει να γίνουν. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με ζητήματα που δεν αφορούν πραγματικά ούτε τους πολίτες ούτε το μέρο των μεταφορών. Πρωτού δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε και αυτοκριτική. Μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειά, πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση και να δούμε τι χρειαζόμαστε, τι δεν χρειαζόμαστε, τι έχει αποβεί χρήσιμο και τι όχι. Και τι δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχει αύξηση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Και υπάρχουν άλλοι κλάδοι στους οποίους έχουν επενδυθεί πολλά κονδύλια για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει συμβεί αυτό και στις μεταφορές. Και αναρωτιέμαι τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και να πω ότι μας μιλάει για βήματα από το 2013 μέχρι το 2015, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο αν δεν έχει γίνει πρώτα το πρώτο στάδιο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και αν δεν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν έχει γίνει. Επίσης, πολύ σωστά αναφέρθηκε ο αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος βλάπτει το περιβάλλον και είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό. Και αυτές οι αναλύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια ελπίζω να μας δείξουν πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, τι θέλει να κάνει η Κομισιόν για να αλλάξει τα πράγματα στο μέλλον. Τώρα έχετε το λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πάρει ό,τι μπορεί από την έκθεση αυτή. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι πραγματικά θεωρούμε εξαιρετικά πολύτιμη τη συνεισφορά σα. Όχι απλώ είναι επίκαιρη, μια και μόλι αρχίσαμε την, ε, την προσπάθεια να βολιδοσκοπήσουμε το που βρισκόμαστε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να δούμε τι έχει ήδη γίνει και τι δεν έχει πάει καλά, τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Σε μια τέτοια προσπάθεια, και αυτό νομίζω ότι προσπαθούσε και ο Επίτροπος να σας ε, πει σε πολλές περιστάσεις, είναι ότι δεν θέλουμε να επινοήσουμε ξανά όλη τη διαδικτύωση των μεταφορών. Αλλά δεν θέλουμε να πετάξουμε και το μωρό με το μωρό του μπάνιου. Δεν θέλουμε λοιπόν να πετάξουμε το μωρό μαζί με το νερό που το κάναμε μπάνιο. Πρέπει να παραμείνουμε όμως ε, πιστοί στις σημαντικές αρχές μας, όπως την κινητικότητα, την διευκόλυνση της κινητικότητας, και την βιώσιμη κινητικότητα. Πρέπει να παραμείνουμε σε κάποιες προτεραιότητες για την πολιτική μεταφορών, δηλαδή την εσωτερική αγορά. Είναι χαρά μου που άκουσα τόσους συναδέλφους σήμερα εδώ να εκφράζονται υπέρ αυτής της καθοριστικής αρχής να μην περάσουμε σε πολλές νέες λεπτομέρειες ή αλλά να εδραιώσουμε όσα ήδη υπάρχουν και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τους καταλληλότερους τρόπους υλοποίησης των ισχυόντων κανόνων. Είναι πολλά τα στοιχεία που προέκυψαν στη σημερινή συζήτηση και θα θέλαμε να τα επεξεργαστούμε προφανώς κι άλλο μαζί σας. Το πλέον σημαντικό νομίζω είναι αυτό που ε, αξιοποίησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σύνθημα. Η διάσταση των ανθρώπων πρέπει να κάνουμε περισσότερα από την πλευρά του χρήστη. Ακόμη και κάποια δουλειά επί της συμπεριφοράς των χρηστών, το σημειώνω αυτό που υπόθηκε, αλλά η διάσταση των ανθρώπων αφορά και τους εργαζομένους, την ποιότητα της εργασίας, τις ευκαιρίες που τους δίνουμε και τη νέα έμφαση, την, την έμφαση που να δώσουμε στις νέες γενιές. Αυτό επιδιώξαμε αρχικά με τη Λευκή Βίβλο. Χρειαζόμαστε μια περισσότερο κοινωνική προσέγγιση στην πολιτική μεταφορών. Έπειτα για τις απογοητεύσεις, ε, την απογοητεύση που χάσετε κάποιοι από εσά, για το πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη χρήση των καυσίμων, γίνεται με πολύ αργό τρόπο αυτό. Όντως, Είχαν ήδη γίνει προτάσει στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο να πάμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε και από την πλευρά τη ενεργειακή αποδοτικότητα σίγουρα πρέπει να τα πάμε πολύ καλύτερα. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι έχουμε ότι έχουμε μια πολύ ναι, καλή νέα προσέγγιση με την Ενεργειακή Ένωση και πιστεύουμε ότι στα θεμέλια αυτά θα μπορέσουμε να χτίσουμε και στο μέλλον ως προς τις υποδομές. Σημειώνουμε όσα λέτε, όντω είναι κρίσιμο θέμα. Επικεντρωνόμαστε στις νέες υποδομές, όχι μόνο στη συντήρηση, αλλά και την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών. Οπότε και αυτές οι επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες. Επίσης, νέα προσοχή δίνεται στις νέες πηγές χρηματοδότησης. Αυτές γίνονται με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χθε είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για το ΕΦΣΥ Ίσως να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά ίσως να χρειάζονται και νέοι τρόποι χρηματοδότησης μέσω της καλύτερης τιμολόγησης της χρήσης των υποδομών. Και όπως τονίσατε κάποιοι από εσά, χρειάζεται και καλύτερη τιμολόγηση των εξωτερικών αναγκών που δημιουργούν ε, οι μεταφορές και τα μέσα μεταφορών. Όλα αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας για να έχουμε μια καλή και αποδοτική πολιτική ε, μεταφορών και ένα τέτοιο σύστημα. Τέταρτη διάσταση, η αλυσίδα της ε, οργάνωσής μας στα διοικητικά και στη διοργάνωση, εδώ πρέπει να δούμε τους βασικούς φορείς που εμπλέκονται. Ε, το ανέφεραν τρία τουλάχιστον από τα μέλη εδώ για τα λιμάνια. Τα λιμάνια έχουν πολύ μεγάλη σημασία ως ένα κομβικό σημείο της αλυσίδας για την ε, σωστή διασύνδεση. Και μετά η αλλαγή της βιομηχανικής μας βάσης. Πρέπει να, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση στις ε, συνθήκες εργασίας, κάτι που μας οδηγεί να δούμε με νέο βλέμμα και την πολιτική ανταγωνισμού και την εμπορική μας πολιτική. Έπειτα, να μην ξεχάσω την επιτάχυνση της καινοτομίας, είναι πολλοί οι βουλευτές που μίλησαν για τη δραστική ε, μετατόπιση προς νέες υπηρεσίες. Εδώ χρειάζονται πραγματικά μεγάλες αλλαγές για να προσαρμόσουμε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην ε, δημιουργήσουμε δυσκολίες στην καινοτομία αλλά να διευκολύνουμε και να επιτρέψουμε να υπάρχουν ισότιμοι κανόνες μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων και φορέων. Εδώ λοιπόν καλό είναι να υπάρχει ε, ισότιμη πρόσβαση ε, για την διάσταση των αστικών κέντρων. Πολλοί από εσά τονίσατε ότι η παράμετρος αυτή των αστικών κέντρων είναι σημαντική. Γι' αυτό και θα περιμένουμε και τη δική σας έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με ανυπομονησία για την αστική κινητικότητα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο εισηγητής έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η σημαντικότερη λέξη που ακούστηκε σήμερα ήταν να μην είναι φλίαρο και κενό το έγγραφο. Γουίσι Wishy-washy που είπε κάποιος. Όμως μπορεί να αποκτούν και απόψε ένα τέτοιο έγγραφο. Από το ECR είπε ένα συνάδελφο που δεν είναι όμω τώρα εδώ, είπε ότι είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και πρέπει να τα δούμε πιο ε, ψύχρεμα. Ο συνάδελφο Ντέλη λέει να είμαι ρεαλιστή. Όταν ε, θέλω να μιλήσω για την πολιτική μεταφορά στην Ευρώπη. Με τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζει έρχεται αντιμέτωπο ένα εισηγητή όταν ε, πρέπει να καταρτήσει μέχρι τον κύριο Άικχαουτ. Σίγουρα η βιωσιμότητα είναι πρόκληση. Και για την καινοτομία και για τη βιομηχανία και για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Θέλω όμω να επιστήσω την προσοχή σα και σε ένα άλλο στοιχείο. Για πολλού το να έχουν αυτοκίνητο είναι και, σημαίνει και χειραφέτηση ως Ευρωπαίοι, Δυτικοευρωπαίοι κυρίως, ε, λέμε ότι ναι πρέπει να είναι, είναι δημόσια αγαθό αυτό και τα λοιπά. Όμως αυτό που είπε η κυρία Μπιλπάο με εντυπωσίασε και πρέπει πράγματι να το λάβω υπόψη. Το είπε και ο συνάδελφος Ερτούκ, ότι η υπότιτλη μεταφορά σε μεγάλο βαθμό απορρέεται από τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, πολλές φορές ε, αποτυγχάνει αυτή η φιλοδοξία στα κράτη-μέλη, προσκρούει εκεί. Για να ολοκληρώσω. Και με τον Γκέτε, είμαστε δύο μήκος κύματος. Αλλά δεν ήταν εύκολο για μένα και για το προσωπικό μου να συνοψίσω μέσα σε ένα έγγραφο όλη την πολιτική μεταφορών. Σίγουρα δεν μπορούσε να είναι τόσο μακροσκελές το έγγραφο για να τα καλύψει όλα. Θα σταλεί προς μετάφραση λοιπόν την επόμενη εβδομάδα και περιμένω ήδη να έχουμε την επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να σας το μεταφράσω εγώ το τσιτάτο του Γκέτε πιο απλά. Το λιγότερο είναι και καλύτερο. Ας προχωρήσουμε όμως. 13 και 14 Απριλίου η παρουσίαση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών 20 Απριλίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 28 Μαΐου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2015. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο διαδικασίε και πρακτικές όσον αφορά τις ακροάσεις των επιτρόπων. Διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τη διαδικασία του 2014. Εγώ είμαι εισηγητή. Και ίσως να θυμάστε ότι δεν ήμασταν και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με, τα, με το γεγονός ότι άλλαξε το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Σεύκοβιτ. Στείλαμε και μία επιστολή στον πρόεδρο Γιούνκερ. Μέχρι τώρα όμω δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Μετά έστειλα και μία επιστολή στον πρόεδρο Σούλτ. Πάλι δεν έλαβα καμία απάντηση. Μόνο ότι ελήφθη η επιστολή. Περίμενα όμω πολύ περισσότερα. Τώρα αποφασίσαμε να συντάξουμε μία έκθεση έτσι ώστε να τοποθετηθούμε για το τι μπορεί να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, αν θέλετε να μιλήσετε, αποχωρήστε από την αίθουσα. Υπήρχε λοιπόν ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ το έργο μας σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογία ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό συνδέεται και με άλλα προβλήματα που απορρέουν από αυτό. Επίσης αναφέρεται στην έκθεση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει από εδώ και στο εξή να ορίζουν δύο υποψήφιους, ένας εκ των οποίων να είναι οπωσδήποτε γυναίκα. Επίσης, η 1η Νοεμβρίου ως ημερομηνία σύστασης της νέας Επιτροπής ε, θεωρώ πως ε, δεν επαρκεί. Θα χρειάζεται, πιστεύω, ένας μήνας παραπάνω, 1η Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος ε, χρόνος και να μην έχουμε τόση πίεση. Επίσης γίνονται αναφορές σχετικά με την διαδικασία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Επιτρόπου Μπούλτ, η οποία το έμαθε τέσσερις ε, μέρες πριν και είχε μόνο τέσσερις μέρες επόμενος χρόνο να προετοιμαστεί για την ακρόαση. Αυτό δεν ήταν δίκαιο ούτε για εμάς ούτε για εκείνη. Δεν ήταν δίκαιη λοιπόν η διαδικασία και πιστεύω πως πρέπει να γίνουν αλλαγές σε αυτό και επίσης η διάσκεψη των Προέδρων αποφάνθηκε για το πώς θα είναι η διαδικασία στο μέλλον. Συμφωνήσαμε λοιπόν για κάποια πράγματα και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τελείως διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω πως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα δικαιώματα συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βιμ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ως Επιτροπή Μεταφόρων. Είναι καλό να τα δούμε αυτά γραπτός. Έχω εκπώνεις και εγώ να εγγραφώ Δεν είναι θέμα μόνο σε Εύκοβιτς, Μπούλτς, γενικά για το φαινόμενο αυτό και για το τι συμβαίνει. Περί αυτού πρόκειται. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι την επόμενη φορά τα ίδια λάθη θα κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα. Είναι στο σύστημα. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις, έχουμε γυναίκες, άνδρες, ε, τη δεξιά την αριστερά, τους κεντρώους. Και θα πρέπει σίγουρα να αντλήσουμε διδάγματα από αυτά τα έγγραφα, να περιορίσουμε τα ασφάλματα που διαπράττουμε, αλλά σε ό,τι αφορά ε, τον ορισμό της Επιτροπής, ε, πιστεύω ότι θα προκύψουν ασφάλματα και στο μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι το ΕΛΚ ζητά να εφαρμόζεται η αρχή ΔΕΟΝΤ. Γνωρίζω ότι επιθυμεί να δίδεται το λόγος και στις μικρές ομάδες, αλλά στις ακροάσεις ε, ένα άτομο από την υποτική ομάδα μπορούσε να μιλήσει τρεις φορές. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία. Θα μπορούσατε να το αναφέρετε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζάκη Φώστερ έχει το λόγο. Ε, θα είμαι σύντομη κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς πιστεύω πως πολύ σωστά τέθηκε αυτό το θέμα υπό συζήτηση, διότι η Επιτροπή Μεταφορών ήταν αυτή που έμεινε ξεκρέμαστη και ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι, κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει ότι δεν είστε αρκετά σαφείς. Όπως και να έχει, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ούτε ήταν δίκαιο για τους ε, οριστείς επιτρόπους. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε προχωρήσει σε μια άλλη διαδικασία, διότι πιστεύω πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της κυρίας Μπούλτ ήταν απαράδεκτη. Είχε μόνο τρεις-τέσσερις μέρες χρόνο να προετοιμαστεί για ακρόαση επιτροπής. Και αυτό πιστεύω πως ε, δημιουργεί προβλήματα και στις δύο πλευρές. Πιστεύω πως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια πρόταση του κράτους μέλους να ορίσει έναν υποψήφιο επίτροπο και χρειάζεται περισσότερη προεργασία προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο του ορισμού ενός υποψηφίου. Εντάξει, εκτός εάν κάποιος ε, πεθάνει ξαφνικά, που δεν το εύχομαι φυσικά σε κανέναν. Τώρα, συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Βάντεκαμπ σχετικά με το ότι υπήρχαν ορισμένοι σε κάποιες επιτροπές που μιλούσαν συνέχεια και δεν άφηναν κάποιους άλλους να τοποθετηθούν. Πιστεύω πως υπάρχει η ανάγκη να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά διότι αντικαθιστώ τον κύριο Τέλος Καπός και Όδη συγγήτρια και μια και τα σχόλιά του είναι στα αγγλικά θα μιλήσω και εγώ αγγλικά. Μπορώ λοιπόν να πω ότι θεωρώ και την έκθεση και το σχέδιο αυτό πλήρες και σκιαγραφεί πιστεύω τα πιο σημαντικά σημεία. Συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 1 για μία προθεσμία σε περίπτωση όπου έχει απορριφθεί ένα υποψήφιος επίτροπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης συμφωνώ με την παράγραφο 4. Η γνώμη μου διαφέρει κάπως όσον αφορά την παράγραφο 2, διότι ναι, μεν ο υποψήφιο επίτροπος θα πρέπει να έχει την τις ακατάλληλες δυνατότητες, αλλά δεν πρέπει να υπαγορεύεται στα κράτη-μέλη το ποιον θα ορίσουν επίτροπο. Σύμφωνοι, είναι πολύ καλή η εξισορρόπηση ανδρών και γυναικών, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εδώ θα ήθελα να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο και να πω ότι θα μπορούσαν να είναι δύο γυναίκες υποψήφοι επίτροποι. Όπως και να έχει όμως, ο πρόεδρος Γιούγκερ θα πρέπει να χαίρεται για το ότι υπάρχουν φιλελεύθεροι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά δεν θα είχαμε τόσες πολλές γυναίκες επιτρόπους. Τώρα, έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το ρόλο της διάσκεψης των προέδρεων και μου λείπει κάπως μία αναφορά στις προτεραιότητες τα προγράμματα του κάθε επιτρόπου. Σε γενικέ γραμμές όμως είμαι ευχαριστημένος και θα υποβάλω μόνο λίγες τροπολογίες οι οποίε θα έχουν σχέση με τα σημεία που μόλις ανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μπρούνο Γκόλνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου το επιτρέπετε, Θα ήθελα να περάσω από το θέμα των ακράσεων των επιτρόπων ε, στη σημερινή μερική διάταξη. Βλέπω ότι προβλέπεται ακρόαση της Επιτρόπου Μπούλτ, που περιορίζεται όμως αδρία των συντονιστών, δηλαδή θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αν δούμε την προηγούμενη ομολογία, σημαίνει ότι οι μη εγγεγραμμένοι πρέπει να ε, εξέλθουν σε αυθούσεις, να εκδιωχθούν από την αίθουσα. Πρέπει να έχουμε μια συζήτηση, όχι με ταξίμον, αλλά γενικά στο Κοινοβούλιο, με τις αρχές του Κοινοβουλίου, για να δούμε αν οι τρεις μη εγγεγραμμένοι μπορούμε ή όχι να εκπροσωπούμαστε, ε, να έχουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Αλλά όταν μιλάμε για ακρόαση, όταν ασχολείται με διοικητικά εντάξει η συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά γιατί όταν έχουμε ακρόαση μιας επιτρόπου να αποκλείονται από την ακρόαση οι μη εγγεγραμμένοι. Αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, και μας στηρεί τη δυνατότητα και εμείς να ασκήσουμε τον έλεγχό μας ε, στο εκτελεστικό σώμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερέστατη αναφορά στη δική μου έκθεση. Τώρα, όταν θα έρθει η κυρία Μπούλ, θα γίνει κάποια ακρόαση, θα συζητήσουμε μία έκθεση και οι συντονιστές το γνωρίζουν αυτό. Εσείς δεν έχετε συντονιστεί διότι δεν ανήκετε σε κάποια πολιτική ομάδα. Και αυτό είναι και ο γενικός κανόνας σε όλες τις επιτροπές. Η γραμματεία των μη εγγεγραμμένων συμμετέχει στην ακρόαση και μετά ενημερώνει. Όμω, οι μία και γραμμένοι, ε, ακριβώ επειδή δεν ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα, δεν μπορούν να έχουν συντονιστεί. Κατ' εξαίρεση θα σας δώσω ξανά το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εντελώς ε, έκτακτο. Πρώτη φορά συμβαίνει. 30 χρόνια με βουλευτή ε, Ποτέ δεν ξαναείδα να είναι δυνατό να παρίστανται συνεργάτες, βοηθοί, αλλά όχι βουλευτές. Μου φαίνεται απίστευτο. Λέτε εσείς ότι μπορείτε ίσως να παραστείτε χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε. Και αυτό συζητείτε βέβαια και μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Αλλά έστω το να μας λέτε ότι δεν μπορείτε καν να ακούσετε εσείς αλλά μπορούν οι βοηθοί σας και έτσι τηρείτε ισότητα, συγγνώμη αλλά με όλο το σεβασμό που τρέφω προς το πρόσωπο και προς το λειτουργήμά σας κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι αυτό είναι κοροϊδία. Εντάξει, κατανοώ πως δεν μπορείτε να το δεχτείτε, δεν μπορεί όμως να αλλάξει τίποτα. Είναι μία απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ακόμα και η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών έχει πιο πολύ συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις, όμως εγώ προσωπικά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάποια εξαίρεση, διότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Τώρα, να πω σύντομα ότι φυσικά θα χαρώ να λάβω τις ετροπολογίες σας. Να σας πω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 5η 19 Μαρτίου, 14 Απριλίου ψηφοφορία στη στην Επιτροπή Μεταφορών, 15 Μαΐου στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και Ολομέλεια τον Μάιο του 2015. Περνάμε λοιπόν με αυτό στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κυρία Τεάντα που θα κάνει την παρουσίαση είναι εδώ. Με χαρά μας σας καλωσορίζουμε λοιπόν για να μας δώσετε μια σύντομη παρουσίαση και τροφή και συζήτηση. Διότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα να συζητήσουμε και πιστεύω πως το ξέρετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας και σας δίνω αυτή αμέσως το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέψατε να έρθουμε εδώ για αυτή την παρουσίαση δεν ονομάζομαι, μου ζητήθηκε να δώσω μια παρουσίαση για τον κατάπλου και και πώς γίνεται η αξιολόγησή μας. Έχω δίπλα μου την συνάδελφο η οποία παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν αν έχετε ερωτήσεις μετά την παρουσίασή μου, η συνάδελφός μου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το θέμα. Το τι κάνουμε λοιπόν σε σχέση με, τη, με τον τομέα των μεταφορών και τη δανειοδότηση. Η ΕΤΕ προσπαθεί να υλοποιήσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών για τρεις βασικούς τομείς. Την ανάπτυξη και την απασχόληση, για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θέλουμε να στηρίξουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την δράση μας για το κλίμα. Θα δείτε στη δεξιά πλευρά την γραφική παράσταση που δείχνει πόσο σημαντική είναι η δανειοδότηση για τον τομέα των μεταφορών. Να δείτε τη συνολική χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΤΕ. Είναι το 20-25% της συνολικής μας δανειοδότησης. Και γι' αυτό υπάρχουν σοβαροί λόγοι Πρώτα απ' όλα τα έργα μεταφορών είναι μακροπρόθεσμα και εμείς ακριβώς παρέχουμε την μακροπρόθεσμη δανειοδότηση, δάνεια μεγάλης διάρκειας. Βιάστηκα λίγο. Ας δούμε τους ε, τομείς για τους οποίους προβλέπουμε στήριξη. Περίπου 50% των ε, δανείων μας πηγαίνουν στους υδροδρόμους και τα έργα των αστικών κέντρων. Την τελευταία δεκαετία έχουμε περίπου 14 δις ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως προς τον τομέα των μεταφορών. Πάνω από το 60% των ε, χρηματοδοτήσεών μας πηγαίνει στη στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων, το βλέπετε και στη γραφική παράσταση, και βεβαίω εδώ υπάρχουν δικημάνσεις στο χρόνο. Βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης, βλέπουμε ότι έγιναν κάπως λιγότερα τα τελευταία δύο χρόνια και είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη δεν προχωρούν τόσο γρήγορα με τα έργα τους. Είναι πολλά τα τεράστια έργα που έχουμε σε εξέλιξη, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και πολλά βέβαια νέα, έχουν, πολύ λιγότερα νέα έχουν αναλυφθεί. Η στήριξη των μεταφορών προχωρά με βάση την πολιτική μας για όπως αποφασίστηκε το 2011 και βεβαίως και βάσει της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής από το 2011 επίσης στις δημόσιες μεταφορές έχουμε δώσει αρκετή έμφαση και έχουμε καλή απόκριση και καλέ αντιδράσει σε αυτήν την πολιτική μας. Τώρα τι προσέγγιση έχουμε αναλάβει σε αυτόν τον τομέα, την ε, διαφοροποίηση των μέσων, την ε, βιώσιμη χρήση των μεταφορών που να είναι φιλική και προς το περιβάλλον, ενώ στην, ε, στις αεροπορικές και οδικές μεταφορές είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Μα περιορίζει το γεγονός ότι στους τομείς αυτούς μπορούμε να χρηματοδοτούμε έργα που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα ή στους τομείς συνοχή. Πέραν αυτών υπάρχουν και συγκεκριμένες απαιτήσει γιατί πρέπει να έχουμε ε, ψηλό οικονομικό κέρδος, ε, αποδόσεις. Συγκεκριμένες απαιτήσει για τους διάφορους επιμέρου τομεί τις προβλέπουμε και τις προβλήματα γιατί δεν μπορούμε να στηρίξουμε όλα τα έργα στα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια για τη στήριξη των οδικών ε, έργων και τις πτυχές ασφάλειας αυτών των οδικών έργων. Βεβαίως φροντίζουμε να υπάρχει συμμόρφωση και με όλες τις ε, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα έργα που χρηματοδοτούμε από την ΕΤΕΦ. Εάν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τη διάσταση των έργων. Νομίζω ε, θα ήταν και για εσάς ενδιαφέρον να το δείτε αυτό. Μας απασχολούν όλες οι φάσεις του κύκλου των έργων, από την αρχή μέχρι την φάση της παρακολούθησης. Πώς αρχίζει να περνάει ένα έργο στον ε, διαβλό μας. Κάποιες φορές έχουμε έτοιμα από τον, ε, από τον υπεύθυνο του έργου, Κάποιες φορές αναθέτουμε εμείς και βλέπουμε ποια έργα θα θέλαμε να προτείνουμε. Αυτό συχνά συμβαίνει στον τομέα των μεταφορών όπου επανειλημμένως έχουμε επευθύνους έργων με τους οποίους ε, εργαζόμαστε συχνά. Μετά, ε, όταν λύθουν τα θέματα της ερεσιμότητας, γιατί δεν είναι όλα επιλέξιμα για να χρηματοδοθούν από την ΕΤΕ, οι έργα στους δρόμους που βλέπετε εδώ, ας πούμε, έξω στην πόλη, δεν είναι κάτι που θα χρηματοδοτούσε η ΕΤΕ, αυτό, αφού περάσει από τον πρώτο έλεγχο, αποστέλλεται στην υπεύθυνη υπηρεσία, υπάρχουν διαβουλεύσεις και συζητούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν, τουλάχιστον τρεις υπεύθυνοι, δύο από το Διευθυντήριο των Έργων και ένας από, από την Υπηρεσία Οικονομικών συζητούν με τον υπεύθυνο του έργου. Αν δούμε την οικονομική αιτιολόγηση, είναι σημαντικό για μας τα έργα που χρηματοδοτούμε να είναι βιώσιμα και τελικώς να έχουν ωφέλη συνολικά για την κοινωνία. τα κοιτάζει λοιπόν η ομάδα μας και βλέπουμε τη διάσταση των ε, διαγωνισμών, του περιβάλλοντος και την κοινωνική έπειτα εξετάζουμε την δυνατότητα του, του εργολάβου, τη δυνατότητα του εργολάβου να φέρει πέρα στο έργο. Και βλέπουμε κατά πόσον το έργο μπορεί να φτάσει στις τελικές φάσεις. Μόλις αρχίζουμε να συζητούμε με τον εργολάβο λοιπόν, βλέπουμε ότι τεχνική βοήθεια θα χρειαστεί για να μπορέσει το έργο να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επί της ουσίας προσπαθούμε να αποτιμήσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να ενέχουν τα έργα, προσπαθούμε να προβλέψουμε παράγοντες όπως τεχνική βοήθεια για να βοηθήσουμε τους εργολάβους να φέρουν εις πέρα στα έργα και ε, ασχολούμαστε και με το θέμα των ε, συμβάσεων, ε, ώστε κάποιες προϋποθέσεις να μας βοηθούν να περατώνονται τα έργα έτσι όπως το θέλουμε εμείς. Ταυτόχρονα, κοιτάζουμε και την πίστοση. Και αν μας ικανοποιεί η δυνατότητα, ε, το συζητούμε με την Υπηρεσία Οικονομικών και ύστερα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον συμβεί αυτό, εγκρίνουμε το δάνειο και αρχίζει η φάση τη παρακολούθηση. Όπω θα φαντάζεστε, η φάση παρακολούθηση για τα έργα μεταφορών μπορεί να είναι και πολύ μακροχρόνια. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της παρακολούθησης των έργων, ε, ανεξάρτητη αποτίμηση, με εμπειρογνώμονες που εργάζονται μόνο στον τομέα των μεταφορών. Όμως και μηχανικοί και οικονομολόγοι μπορεί να μπλέκονται εδώ, παντού που έχουμε εντολή. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για την ΕΤΕ και έχουν ε, γνώσεις για το θέμα αυτό. Έχουν συνηθίσει να εξετάζουν έργα και μάλιστα σε διαφορετικέ χώρες. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω έχει τεθεί ένα θέμα για το αν θα κάνουμε την ίδια αποτίμηση για όλα τα έργα που θα προτείνονται και ε, για την ώρα αυτό συμβαίνει. Και τα έργα που προωθούμε και τα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν με το ΕΨΙ. Θα δίνουμε την ίδια προσοχή. Με τη δέουσα προσοχή εξετάζουμε τις βελτίστες πρακτικές και κοιτάζουμε αυτές να ε, υπάρχουν και στην περιπτώση των έργων που χρηματοδοτούμε. Και μας ενδιαφέρει και το, το αμοιβαίο όφελος των έργων. Έχουμε βάσει δεδομένων με δειγματοληψία για το κόστος και έχουμε βέβαια συνηθίσει να κοιτάζουμε τέτοια έργα με βασικούς αριθμούς αναφοράς τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Πολύ συχνά οι εργολάβοι είναι πολύ αισιόδοξοι, υπεραισιόδοξοι μάλιστα για τα έργα τους και πολλές φορές είναι και προκατελημένοι στις αριθμιστικές τους προβλέψεις. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο να κατεβάζουμε κάπως τα αισιόδοξα αυτά όρια που έχουν προβλέψει και να τους επαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μέρος των διαφόρων μοντέλων που έχουμε ε, κατασκευάσει με το αμοιβαίο, με την ανάλυση του αμοιβαίου, με την ανάλυση του κόστους ωφελίας. Και βλέπουμε κατά πόσον η ζήτηση για το έργο μπορεί να μας οδηγήσει στην απαραίτητη επιτυχία. Κοιτάζουμε την ε, ανάλυση κόστους ωφελίας και το κατά πόσον το αποτύπωμα του έργου θα είναι αυτό που θέλουμε. Βλέπουμε τι γίνεται και με το περιοδική λοιπόν διάσταση, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και το άλλο μπορεί να περιλαμβάνει η ανάλυση κόστους ωφελίας. Πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΕ έχει και μια στρατηγική για το κλίμα που έχει περάσει και από δημόσιες διαβουλεύσεις. Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει, γιατί ο τομέας των μεταφορών είναι ένας τομέας μεγάλος και σημαντικός και, και από αυτή την άποψη. Ως προς το screening των έργων, έχουμε μία μεθοδολογία της προστιθέμενης αξίας όπως την έχουμε ονομάσει. Αυτή η μεθοδολογία βάσει των ε, βέλτιστων πρακτικών και πολλές, πολλά ιδρύματα έχουν το ίδιο σύστημα. Ε, αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα του έργου, δηλαδή η βαθμολόγηση του κατά πόσο είναι ποιοτικό. Δεύτερον, κατά πόσον έχει ε, επιτυχία προς το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο αυτό. Και τρίτον, ποια είναι η συμβολή της ΕΤΕ στο έργο. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου βαθμολογούμε τα έργα. Και βάσει αυτού των των ε, κλιμάκων αποφασίζουμε τι αποτέλεσμα θα δώσουμε στα έργα αυτά. Έχουμε τα βασικά αποτελέσματα, τα ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα και την απόδοση των έργων. Να σας δείξω ένα παράδειγμα, τι έγινε πέρσι με τέτοιου είδους έργα. Βλέπετε ότι τους δείκτες μας τους χρησιμοποιήσαμε και για την προβολή ενός έργου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται και για τη μέτρηση, αλλά και για να δούμε τι αποτέλεσμα πετύχαμε σε σχέση με αυτό που βλέπαμε και για το κατά πόσο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και σε νέα έργα. Προσπαθούμε δηλαδή να διδαχθούμε από, προγράμματα που έχουν, από έργα που έχουν ολοκληρωθεί στο παρελθόν. Μερικά παραδείγματα πρωτού ολοκληρώσω. Μεγάλη προτεραιότητα για τα έργα. Βλέπετε να δίνετε και στις εικόνες στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ένα έργο του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου στην Ισπανία, λόγω χάρη, ε, στην εικόνα έχω ένα έργο επίσης που πέρασε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο, το έργο κινητικότητας για το Λονδίνο, η στήριξη των αυτοκινητών δρόμων, των θαλάσσιων δρόμων και ένα περσινό έργο που αφορούσε σκάφη και αναβάθμιση σκαφών με, με χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου και αντικατάσταση των κινητήρων τους. Αυτό σας δίνει μερικά παραδείγματα και κάποια συμπεράσματα για να ολοκληρώσω ποιε είναι οι τάσει που επικρατούν στην ΕΤΕ από την θέσπιση της πολιτικής μα για τι μεταφορέ το 2011 βλέπουμε να είναι πρασινότερη η προσέγγιση μα, Δηλαδή το θεματολόγιο, το χαρτοφυλάκιό μα έχει εμπλουτιστεί σε σχέση με τι οδικέ και αεροπορικέ μεταφορέ που ισχύει τώρα. Και για το μέλλον τη επιλογή έργων Βεβαίω έμφαση θα υπάρχει να έχουμε αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά δίκτυα από τα πολλά, αλλά ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε μερικά κράτη-μέλη που χρειάζονται να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα δίκτυα που θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν καλύτερα και που πρέπει να εφαρμόσουν ευφιέστερες λύσεις κινητικότητας ή ολοκληρωμένες. Βεβαίως το ERTMS παραμένει ένα σημαντικότατο μέρος των ε, έργων μας και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον κατά την υλοποίηση των νέων, ε, επενδύσεων για τις ε, συνδρομικές μεταφορές. Μας ενδιαφέρουν και οι νέες ιδέες όπως η ηλεκτροκινικότητα ή οι εναλλακτικές τα εναλλακτικά καύσιμα. Δεν έχουμε ακόμα πολλά τέτοια έργα, αλλά θα προχωρήσουμε ω προ αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον. Θα σοπάσω αφού σα πω και δύο τελευταία λόγια. Ε, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν έχουμε λίγο χρόνο ε, και λιγότερους πόρους, σημαντικό είναι οι πόροι να ε, κατευθύνονται στα καλά έργα, στη σωστή επιλογή. Και αυτό βεβαίω αφορά και την τεχνική διάσταση των έργων. Έμφαση πρέπει να δοθεί και στο συστημικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με τα δημοτικά δίκτυα. Και νομίζω ότι εδώ ο σχεδιασμό του πλαισίου μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχω δει σε άλλη μέρα του κόσμου. Ένα λοιπόν σαφές μήνυμα ισχύει όταν κανείς προτείνει πράγματα σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι πρέπει τα έργα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε ως δι. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς ένας αυτοκινητόδρομο να χτίζει ένα αυτοκινητόδρομο όταν απλώς μπορεί να καλυφθεί με έναν δρόμο. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας είναι αυτός. Και κάτι ακόμη που βλέπουμε είναι οι εργολάβοι να θέλουν να ολοκληρώσουν το έργο πολύ γρήγορα, αλλά να μην γίνεται σωστά η αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτό μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα τελικά και γι' αυτό, βάσει τι εμπειρίε μα, έχουμε δει ότι ο βέλτιστο σχεδιασμό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Όταν μιλάμε για επενδύσει σε μεγάλε υποδομέ και σχετικά έργα. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα έργα είναι μεγάλες διάρκειες και ότι βεβαίως είναι και βιώσιμα. Με αυτά και με αυτά να σας ευχαριστήσω ξανά που μας καλέσατε σήμερα και ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε. Yeah, thank you very much as well. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Ο κύριος Βάντεκαμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος πως θα θέλει και ο συνάδελφος Πίπερ να μιλήσει. Να πω ότι το θετικό που άκουσα από εσάς είναι ότι τα τελευταία χρόνια στους σιδηροδρόμους έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις και στη συντήρηση. Τώρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητιέται αρκετά η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πιστεύω πως ε, δεν είναι ανάγκη να σας κάνω μία περίπλοκη ερώτηση, αλλά εσείς πώς εκτιμάτε την δουλειά που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα. Και κάτι άλλο, οι διασυνοριακές απόψεις. Υπάρχουν για παράδειγμα διασυνοριακές οδοί, υπάρχουν όμως και ποδηλατόδρομοι π.χ. στο Λονδίνο οι οποίοι δεν είναι διασυνοριακοί. Εδώ υπάρχει θέμα επικουρικότητας του Connecting Europe και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό. Και κάτι άλλο, η διασύνδεση των διάφορων μέσων μεταφοράς και των διάφορων μέσων χρηματοδότησης. Υπάρχει η ΕΤΕ, υπάρχει το ΣΕΦ, υπάρχουν τα δημόσια κονδύλια και οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης, για παράδειγμα η χρηματοδότηση μέσω cloud. Εσείς Πώς ε, αξιολογείτε αυτούς τους τρόπους χρηματοδότησης, ορισμένες φορές καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ερτούγκ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω και εγώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε έναν εκπρόσωπο της ΕΤΕ σήμερα μαζί μας. Η σημασία του έργου σας έχει αποδειχθεί και τώρα αλλά και γενικότερα. Έχω αρκετές ερωτήσεις, ελπίζω να μην σας κουράσω. Είναι ερωτήσεις όχι δύσκολες, αλλά για την καλύτερη κατανόηση του έργου σας. Μας αναφέρατε την ανάπτυξη. Και τους, ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τους ε, ανάδοχους. Έπειτα μας αναφέρατε την προστιθέμενη αξία ως μέθοδο που ακολουθείτε και αυτήν την αξιολόγηση. Υπάρχει μία συμβατότητα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία συνυπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση, τουλάχιστον αυτή η διαλογή σε προγενέστερο στάδιο. Υπάρχει σύστημα πόντων, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείτε και εάν ναι, πώς αξιολογείτε εσείς ε, αυτούς τους πόντους, πώς δίνετε πόντους και ποια κριτήρια είναι αυτά που χρησιμοποιείτε για να αξιολογήσετε λοιπόν σε αυτό το προγενέστερο στάδιο τα προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσετε. Έπειτα αυτή η πράσινη προσέγγιση στην Ασυπλού είναι κάτι που με χαροποίησε πάρα πολύ καθώς και η συμπερίληψη του αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα. Είναι και αυτό μία άποψη η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί και να διατηρηθεί τουλάχιστον στην επιλογή των προγραμμάτων. Έχω και μία ερώτηση παρόμοια με εκείνη του συνάδελφου Βάντεκαμπ. Έχουμε ακούσει πολλές λέξεις κλειδιά. Δάνεια από την ΕΤΕ, επιχορηγήσεις, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπερίληψη ιδιωτικών επενδυτών και τα ομόλογα έργου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα όλους αυτούς τους τρόπους χρηματοδότησης. Θα ήθελα να το μάθω αυτό για να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο που εργάζεστε. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, η προσφορά των υπηρεσιών σας δεν ισχύει για νέες κατασκευές, αλλά για συντήρηση και ανακατασκευή. Διακόπτει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, αν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ να περάξετε έξω, γιατί διακόπτεται τη συζήτηση. Τώρα, εάν εγώ, για παράδειγμα, θέλω να κάνω μία συντήρηση ή μία επέκταση, μία μετασκευή κάποιου προγράμματος και είμαι ανάδοχος ενός έργου. Θα λάβω χρηματοδότηση μόνο για συντηρήσεις και για ανακαινήσεις ή και για καινούργια προγράμματα. Και επίσης, ποιο είναι το δικό σας ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του κόστους ενός έργου. Για παράδειγμα, αν κάτι κοστίζει 70 εκατομμύρια. Ποια είναι η δική σας συμμετοχή, ποια είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και αν υπάρχουν κάποια κενά, από πού καλύπτονται, ποιος τα χρηματοδοτεί και ποιο είναι το ανώτατο όριο του ποσοστού συμμετοχή σας. Και τι γίνεται στην περίπτωση χρηματοδότησης έργων σε τρίτες χώρες. Πολλές ερωτήσεις έχω, το ξέρω και ελπίζω να μην σας κουράσουν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όταν κάποιος κάνει πολλές ερωτήσεις, συνήθως καλύπτει και τους επόμενους ομιλητές. Πιστεύω πως ε, μας βοήθησε πάρα πολύ η παρουσίασή σας. Ε, αλλά να πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για τα κριτήρια και αυτό που για μας είναι πολύ σημαντικό, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δεν ήταν ε, εξίσου σημαντικό για σας. Ήταν όχι στην πρώτη θέση των ε, προτεραιοτήτων σας και μου έκανα κάποια εντύπωση αυτό. Επίσης μας είπατε για κάποια αστικά ε, έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται μόνο όταν βελτιώνουν την κινητικότητα. Επίσης είπατε ότι θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία για όλα τα έργα. Αυτό ισχύει, διότι στην περίπτωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και του ΣΕΦ υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται. Και από ό,τι έχω καταλάβει, στα πλαίσια του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει οι ιδιωτικοί επενδυτές να είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε πρώτο στάδιο. Και τέλος, πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο και πρέπει να φύγω, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω πριν δώσετε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, τουλάχιστον μας ειδοποιήσατε. Κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις, δύο συγκεκριμένα για εσάς. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε ιδιωτικούς επενδυτές να επενδύσουν το μεταμεταφορών. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φυτρώνει στα δέντρα το δημόσιο χρήμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις για τα διάφορα έργα επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Μάισνερ όταν μίλησε για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Οι μεταφορές, κατά την άποψή σα δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη δυνητικά. Καρή Μαντελή τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Διευθύντρια για την παρουσίαση. Έχω πολλά ερωτήματα και διευκρινήσεις ε, θα ήθελα για διάφορα πράγματα. Είπατε ότι συγχρηματοδοτείται βιώσιμα έργα. Εδώ είμαι, εδώ. Καλημέρα. Αυτή η βιωσιμότητα, εσείς είπατε κάποια κριτήρια για αυτήν. Σήμερα θα ήθελα να μου πείτε όμως αν η ΕΤΕ είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει τα κριτήρια που γνωρίζουμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και στο Connecting Europe Facility και σε ό,τι αφορά το, έργο, το, το πρόγραμμα Juncker. Αυτό είναι το πρώτο μέρο, δηλαδή τα κριτήρια που υπάρχουν ήδη και ισχύουν για αυτά τα δύο προγράμματα, ΣΕΦ και διευρωπαϊκά δίκτυα, είτε για την ευρωπαϊκά ελαχιστοποίηση εξωτερικού κόστους, μείωση κομπών εξαιτία του άνθρακα. Αυτά θα ισχύσουν ή ε, απλά ο σεβασμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θα σεβαστούμε για την ισχύουσα νομοθεσία. Πρώτο ερώτημα και δεύτερο, είστε μέλος και της Επιτροπής Επιλογής των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος ε, Juncker. Δύο ερωτήσεις. Μίλησατε για βιωσιμότητα, επαναλαμβάνω. Τι θα πει αυτό. Τι είναι αυτή η βιωσιμότητα για σας. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένο. Νούμερο. Πόσα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν από το 2009 ως το 2014 στον τομέα των μεταφορών. Ξέρετε, να μας δώσετε έναν αριθμό πραγματικά. Αυτό λοιπόν το στοιχείο θα ήθελα και επόμενο ερώτημα. Πώς θα ενθαρρύνετε τις χώρες οι οποίες σήμερα δυστυχώς δεν λαμβάνουν ε, βοήθεια ε, μιλάω για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως, στον τομέα των υποδομών. Κυρίω για τις ιδεοδρομικέ μεταφορές πώ θα τι βοηθήσει αυτέ τι χώρε και μήπω η ΕΤΕ θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο. Έχουμε ένα, μια σύνοδο κορυφή για το κλίμα, πάρα πολύ σύντομα. Μας περιμένουν να, να είμαστε πρωτοπόροι. Μπορεί να βοηθήσει και η ΕΤΕ για την οικολογική, για αυτόν τον οικολογικό μετασχηματισμό. Όταν μιλάμε επίση για αστική ε, κινητικότητα και συνδυασμού μεταφορές, θα πρέπει να επιλέξουμε τέτοιου είδους έργα και όχι πάρα πολύ μεγάλα ε, φαραωνικά έργα. Και ενώ όλοι το καταλάβατε, Λιόν μπράβο, το καταλάβατε όλοι. Μπορείτε λοιπόν να μου δώσετε τις διευκρινήσεις. Wenn Εάν πραγματικά δεν είχατε κάνει αυτή την ερώτηση, θα αναρωτιόμουν τι συμβαίνει. Αλλά η κυρία Λούνγκραν έχει το λόγο τώρα. Ο κύριος για τη χρηματοδότηση του Connecting Europe Facility. Ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε ότι δίνεται δάνεια με καλή απόδοση, μιλήσατε για 140 δις νομίζω, με το σχέδιο Juncker. Μετακινούμε χρήματα από το ΣΕΦ σε ένα ταμείο επενδύσεων, όπου εκεί υπάρχει ψηλότερο ρίσκο. Έχουμε για τις μεγάλες επενδύσεις αυτό το ταμείο θέλουμε να έχουμε 350 δις. Ξεκινώντας όμως από 20, με ε, αυτό τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα ε, επί 15 ή όμως ο κίνδυνο, ψηλό το ρίσκο. Και θέλουμε εγγύηση από τι τράπεζες νέα Δάν. Άρα για τις τράπεζες καλά είναι τα πράγματα, αλλά μήπως είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο για το πρόγραμμα Juncker. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση σχετικά με τη διαφορετική αξιολόγηση των οδών και των διάφορων άλλων έργων. Καταλαβαίνω ότι για μια υδάτινη οδό ή μια σιδηροδρομική οδό α, περιμένετε λιγότερα έσοδα. Όμως, τι γίνεται σε τεχνικό επίπεδο, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Εντάξει, η απόδοση των ε, χερσαίων οδών είναι κάτι που μπορώ να καταλάβω. Το κέρδος έρχεται από τη χρήση. Στην Γερμανία έχουμε τον αυτοκινητόδρομο 1, τον αυτοκινητόδρομο 7, οι οποίοι στηρίζονται με ευρωπαϊκά ε, κονδύλια και καταλαβαίνω ότι είναι μια κερδοφόρος ε, επιχείρηση, project και για ιδιωτικούς επενδυτές. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση μιας ε, πλωτής οδού. Υπάρχουν λιγότερα έσοδα που αναμένεται ή Πώς μπορείτε να χρηματοδοτήσετε επιπροσθέτως ε, αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι λιγότερο κερδοφόρα για τους ε, ιδιωτικούς επενδυτές. Και πολλές φορές να πω ότι ορισμένα προγράμματα που αφορούν υδάτινες ε, οδούς δεν είναι καθόλου εύκολο να χρηματοδοτηθούν, δεν θεωρούνται κερδοφόρα. Έπειτα, να σταθώ σε κάτι που ρώτησε και ο κύριος Βάντεκαμπ. Το Λονδίνο, μετρό, ανάπτυξη αστική είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω γιατί έχει κάτι τέτοιο ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όταν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και τέλος, να ρωτήσω κάτι για το σχέδιο Juncker και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κάνετε εσείς και σε αυτό που προτίθεται να κάνει το ΕΦΣΥ. Δώστε μας ένα παράδειγμα ίσως για να καταλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ντομινίκ Κρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συντομία, μια παρατήρηση και δύο ερωτήσεις. Η παρατήρησή μου είναι ότι νομίζω ότι είναι καιρός να επαναλάβουμε ότι η ΕΤΕ είναι τράπεζα και όχι κάτι άλλο. Και από αυτή την ιδιότητα επενδύει χρήματα, δεν τα χαρίζει και είναι πολύ διαφορετικό ο ρόλο από ένα πολιτικό όργανο. Η τράπεζα επενδύει με ρίσκο και βέβαια με την ελπίδα ότι θα έχει απόδοση στην επένδυσή της. Αλλά το ρίσκο ε, θέλει να το ζυγίσει έτσι ώστε να έχει και κέρδος στο τέλος. Και η πρόσβαση στην αγορά είναι καλή. Γι' αυτό θέλει καλή αξιολόγηση τράπεζα. Το πρόβλημα των επενδύσεων της ΕΤΕ είναι ότι θα έχει πάντοτε ε, το βλέμμα στραμμένο ε, στην ευρωπαϊκή αξία των έργων και τέθησαν κάποια ερωτήματα και στον κίνδυνο, στο ρίσκο. Και θα πρέπει να τα ζυγίσει αυτά τα δύο ε, για να πάρει τη θετική αρνητική απόφαση αν είναι αποδεκτό το ρίσκο και αν υπάρχει αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή αξία. Δύο ερωτήσεις έχω προς εσάς. Πρώτη ερώτηση. το πλαίσιο των θεσμικών οργάνωσης Ένωσης και από τον έλεγχο της ε, Επιτροπής υπάρχουν ε, τα εγγυητικά εργαλεία, τα ομόλογα έργων παραδείγματο χάρη. Τι σχέσεις εργασίας, ή λειτουργικές σχέσεις θέλετε να έχετε ως ΕΤΕ με αυτά τα ταμεία εγγύησης κινδύνων, ε, κονδύλια που διαχειρίζεται η Κομισιόν και το έψι το Στρα... Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα υπάρχει ανταλλαγή επικοινωνία για αυτά τα θέματα, μεθοδολογικές ανταλλαγές θα υπάρξουν κτλ. Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει η Επιτροπή η επενδυτική που επιλέγει τα σχέδια που θα μπορούσαν να χρηματοδοθούν στο πλαίσιο του ΕΦΣΙ. Και επειδή όμως πρόκειται για τράπεζα, μετά από αυτή την επενδυτική επιτροπή φαντάζομαι ότι το ΔΣ θα αποφασίσει τελικά για αυτά τα έργα. Και εδώ έρχεται το δεύτερο ερώτημα. Ποιο λαμβάνει την απόφαση, η Επενδυτική Επιτροπή, που ορίζεται στην πρόταση κανονισμού τη Κομισιόν, ή το Δικτικό Συμβούλιο τη Τράπεζα τελικά αποφασίζει τι επενδύσει θα γίνουν. Άρα η το δικτικο συμβουλιο τη τραπεζα τελικα αποφασιζει τι επενδυσει θα γινουν αρα επιτροπη ε, επενδύσεων, η Επενδυτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ε, ρόλο ή παίρνει κάποια απόφαση. Ja, jetzt habe ich mich nochmal als letzter Θα πάρω τελευταίο στο λόγο. Φυσικά και όλοι επιθυμούμε την ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ακούστηκαν πάρα πολλέ κριτικέ για το ότι ένα ποδηλατόδρομο ή ένα μετρό σε μια πόλη δεν έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όμω μιλήσατε για ειδικέ προϋποθέσεις και η διασυνοριακή σύνδεση είναι μια αποφασιστική προϋπόθεση. Πρέπει να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κενό 8 χιλιόμετρων στη σιδηροδρομική σύνδεση Γερμανίας-Τσεχίας. Εδώ και 25 χρόνια, παρότι υπάρχουν τα χρήματα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε αυτό το κενό. Όμως, παρομοίως και στη, στα γαλλογερμανικά σύνορα ανάμεσα στο Στρασβούργο και στο Κολμάρ υπάρχει και πάλι κάποιο κενό στην σιδηροδρομική ε, σύνδεση. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα και αυτό οδήγησε στη διακοπή της ε, σιδηροδρομικής συγκοινωνίας και δεν έχει διορθωθεί μέχρι τώρα. Και πραγματικά αυτά είναι αναγκαία ε, προγράμματα έτσι ώστε να αναπτυχθούν ταυτόχρονα και τα δύο κράτη τα οποία αφορά το πρόβλημα. Τώρα, αυτό το project έχει εκτιμηθεί από τη μία πλευρά ότι θα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια και από την άλλη, από την πλευρά της Γαλλίας, ότι θα κοστίσει τα δεκαπλάσια. Αυτά είναι μεγάλα ποσά σίγουρα, όμως υπάρχουν προγράμματα τα οποία κοστίζουν πολύ λιγότερο, τα οποία θα είναι πιο εύκολο να χρηματοδοτηθούν και θα δώσουν ακόμα περισσότερη προστιθέμενη αξία. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, έχετε απορρίψει ποτέ κάποιο πρόγραμμα επειδή δεν ήταν χρηματοδοτήσιμο Σίγουρα όταν κάτι κοστίζει 40 δισεκατομμύρια και είμαι ιδιωτικό επενδυτή, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσω. Όμως, από την εμπειρία μου 30 ετών στον χώρο των μεταφορών, πιστεύω πως η ανάλυση κόστους όφελους είναι κάτι που δεν μας χρησιμεύει πάρα πολύ. Υπάρχει η σύνδεση, για παράδειγμα, Βερολίνου με μια πόλη της Πολωνίας, όπου ε, το κόστος της κατασκευής της έχει εκτιμηθεί ως μη βιώσιμο. Υπάρχει όμως τώρα μια δεύτερη μελέτη η οποία υπολογίζει πολύ μικρότερο κόστος. Εσείς πώς μπορείτε να υπολογίσετε το πραγματικό κόστος. Ε, πιστεύετε τον πρώτο που θα σας ε, κάνει μια μελέτη, πώς το συγκρίνετε αυτό. Κάνετε δικές σας μελέτες, ε, τις αναθέτετε σε ιδιωτικές εταιρείες. Τι κάνετε σε περίπτωση που θέλετε να διαπιστώσετε αν έχει υπάρξει αντικειμενικότητα, αν έχει υπάρξει απάτη. Και τέλος. Αυτή η αύξηση, 15πλάσια αύξηση του σχεδίου Juncker, είναι εφικτή ή είναι ένα όνειρο. Δηλαδή στην αρχή είχαμε 3, μετά τα 3 τα κάναμε 15 και μετά τα 15 τα κάναμε 350. Πώς γίνεται αυτό. Εσείς θεωρείτε πως ε, αυτά τα ποσά είναι ρεαλιστικά, είναι ε, εφικτά βλέπω μηδιάτε. Γι' αυτό σίγουρα θα έχετε κάποια απάντηση να μου δώσετε. Έχετε το λόγο εσείς και η συναδελφό σας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα ερωτήματα και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω τα περισσότερα εξ αυτών. Αλλά καταρχάς να αναφέρω ότι φυσικά και είμαστε στη διάθεσή σας ε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και στο πλαίσιο διμερών ε, επαφών Οπότε μπορούμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία, φυσικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμά. και αυτό και προσπάθουμε να πετύχουμε. Εδώ είμαστε για να προωθήσουμε ευρωπαϊκά έργα και αυτά να υλοποιήσουμε. Ίσως να μην το έγραφα στις διαφάνειες, αλλά είναι και ο λόγος της ύπαρξής μας ουσιαστικά. Το ίδιο ισχύει και για τα διασενοριακά έργα. Πολλά τέτοια ε, έργα συγχρηματοδοτούμε και θέλουμε τους εργολάβους άνθρωπους να τους βοηθήσουμε. Θέλουμε επίσης να υπάρξει και συντονισμός μεταξύ των χωρών. Αυτή είναι η στόχη μας. Η τράπεζα, όπως γνωρίζετε, έχει συγκροτήσει και ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οπότε δίνουμε συμβουλές στους αναδόχους. Τώρα, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφόρων. Φυσικά και αυτή είναι η βασική μας δραστηριότητα και από τα αριθμητικά στοιχεία βλέπετε ότι εκεί επενδύουμε τους περισσότερους πόρους. Ένα έργο που εγκρίθηκε από το ΔΣ την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο. Ε, το επενδύουμε, ε, επενδύουμε σε αυτό γιατί θέλουμε έγκαιρη δράση. Παραδείγματο χάρη για του πολίτε που ζουν στι πόλει. Πολλοί από αυτού ζουν σε πόλει. Θέλουμε δύο Και έχει και ευρωπαϊκό στόχο η επένδυσή μα. Φυσικά τα ευρωπαϊκά δίκτυα όμω είναι η βασική μα προτεραιότητα και τα διευρωπαϊκά και τα διασυνοριακά έργα. Ρωτήσατε. Μεθοδολογία για την προσταμένη αξία. Πράγματι. Ίσως θα άξιζε να το δούμε πιο αναλυτικά. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι να είμαστε όσο να τον πιο αντικειμενικοί ε, στα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και στην αξιολόγηση που κάνουμε. κάνουμε την αξιολόγηση και έπειτα την παρακολουθούμε. Θέλουμε να είναι αντικειμενική αυτή η αξιολόγηση, άρα να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Βλέπουμε μετά τον κύκλο του έργου και αυτό μας δίνει πρώτα απ' όλα. Να κάνουμε πολύ νωρί στο πλαίσιο της δικασίας αποφάσεων τη διαλογή των έργων και επειδή είπε ο πρόεδρος αν κάνουμε διαλογή, φυσικά και κάνουμε διαλογή των έργων. Και αν δεν θεωρούμε ότι είναι βιώσιμα τα έργα ή δεν θα αξιοποιηθούν, δεν τα επιλέγουμε. Γι' αυτό εντάσσεται και στην όλη διαδικασία αποτίμησης, εκτίμησης των έργων. Άρα, πώς μας κάπως να βαθμολογήσουμε αυτά τα έργα με κριτήρια την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Το ίδιο κάνουμε και με την ανάλυση κόστος ωφέλης. Και συμφωνώ πολύ με τα σχόλια που εκφράσατε. Σίγουρα μπορούμε να έχουμε ό,τι αποτελέσματα θέλουμε σε αυτή την ανάλυση κόστος-οφέλους. Έχουμε όμως εσωτερικά ένα εργαλείο, πηγαίνει ο εμπειρογνώμων, εξετάζει πολλά έργα σε πολλές χώρες. Έχουμε βάση δεδομένων, ξέρουμε και το κόστος και πηγαίνουμε συνέχεια επί τόπου και αξιολογούμε την κατάσταση, μιλάμε και με τους εργολάβους. Δεν παίρνουμε απλά τα στοιχεία που μας δίνουν οι εργολάβοι όμως, προσπαθούμε να τα μελετήσουμε και εμείς και να αξιολογήσουμε και να δούμε αν είναι λογικά, λογικές εκτιμήσεις. Νομίζω για τη μεθοδολογία αποτύπωμα άνθρακα επίσης κάτι με ρωτήσατε. να το συζητούμε και με άλλους που ενδιαφέρονται πολύ για αυτή τη μεθοδολογία. Εδώ επιδιώκουμε κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι αυτό θα συνιστά και προσθέμενη εξέ για τους υπεύθυνους λήψη αποφάσεων. Αυτό το κριτήριο, δηλαδή το αποτυπώματος άνθρακα. Να πω επίσης ότι Εργαζόμαστε και με άλλους φορείς. Σπαθούμε να περάσουμε τα μηνύματα και αλλού. Άλλο ερώτημα. Αν χρηματοδοτούμε προγράμματα εκτός Ένωσης, ναι είναι η απάντηση. 10% των δανείων μας είναι εκτός Ένωσης, εκεί όμως που έχουμε ειδική εντολή, βέβαια, είναι πολύπλοκα τα έργα σε ό,τι αφορά την τεχνική ιδέα. επιμήλεια αλλά και με άλλους φορείς ε, όπως είναι η, Διεθνής η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργαζόμαστε. Αν έχουμε την ίδια δέσομελή για έργα αποκατάσταση, ναι έχουμε. Τη συντήρηση δεν την ε, χρηματοδοτούμε βέβαια. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λειτουργικό κόστος. Βελτίωση, συντήρηση ναι είναι επιλέξιμη δραστηριότητα. Παραδείγματο χάρη αναβάθμιση δυναμικού δικτύου στην Νότια Ευρώπη. Έχουμε χρηματοδοτήσει πολλά τέτοια έργα. Και νομίζω ότι τα ωφέλη, το όφελο μάλλον αυτό που προσφέρει η τράπεζα είναι ότι ξεκινάμε διάλογο και χρηματοδοτούμε, χρηματοδοτούμε άλλα πολλά συνδρομικά project στην Νότια Ευρώπη. Έχουμε εμπειρία ετών με αυτούς τους ε, αναδόχους ή εργολάβους και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα προωθήσουμε με λογικό τρόπο αυτά τα έργα και να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες. Δεν χρειάζεται να έχουμε στεδρόμους υψηλής ταχύτητας παντού στην Ευρώπη με τη μια. Μπορούμε να κλιμακώσουμε τις επενδύσεις μας και να τις προσαρμόσουμε εκεί που οι ανάγκες είναι πιο έντονες. Νομίζω ότι... Έγινε μια ερώτηση για το crowdfunding μπορούμε να πάμε στο 50% να καλύψουμε το 50% του κόστου των έργων στον τομέα των μεταφορών ή το 30% ανάλογα με το έργο, εξάρτητα από την κατηγορία του έργου. Ε, Συνήθω ε, τα ποσοστά διαφέρουν, αλλά περίπου φτάνουμε στο 30% χοντρικά. Το όριο είναι 50%. Φτάνουμε στο 50%. Υπήρχε και μια ερώτηση ε, για τους για τις κοινωνικές, για τα κοινωνικά ωφέλη. Δεν έλεγα για επιστροφές λοιπόν οικονομικές αναγκαστικά, αλλά και για την ε, αξία του ίδιου του έργου και το τι ωφέλη μπορεί να αποφέρει για την κοινωνία. Όταν μιλούσα για τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, θα πρέπει να υπάρχει υψηλότερο ποσοστό επιστροφής Και για να είναι ευδιάκριτη η αξία των έργων, θα πρέπει και η οικονομική τους, το οικονομικό κέρδος που αποφέρουν να είναι σαφές. Εδώ πάντως μιλάμε για οικονομικά ωφέλη. Κοιτάζω αν μπορέσω να καλύψω λίγο πολύ τις ερωτήσεις που απευθύνονταν περισσότερο σε μένα. Τώρα για το πακέτο Juncker να δώσω το λόγο στη Μαρία. Σε παρακαλώ Μαρία. Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μαθηκά σε κάποιες ερωτήσεις και να πω το τι είναι η ΕΤΕ. Είμαστε τράπεζα αλλά όχι μόνο τράπεζα. Created by, by the Treaty of Rome. Αλλά και ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο είμαστε. Δεν λειτουργούμε όπως οι υπόλοιπε τράπεζες. Το ακούσαμε από κάποια μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό ότι ε, στις τράπεζες λένε συνήθως είμαι τράπεζα, εμπιστέψουμε. με τους άλλους μπορεί να μην ισχύει αυτό, να είστε καχύποπτοι, αλλά σε εμάς ισχύει. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Αυτό πρέπει να σας πω σήμερα. Επειδή είμαστε τράπεζα, όχι, όντω δεν δίνουμε επιδοτήσει και δεν είμαστε και διάβλο για επιδοτήσει. Δάνεια δίνουμε και περιμένουμε τα δάνειά μα να αποπληρωθούν. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να λειτουργούμε ω κανονική τράπεζα. Δεν δουλεύουμε για το δικό μα το κέρδο. Χρηματοδοτούμε τον εαυτό μα στην αγορά κεφαλαίων από την αγορά κεφαλαίων. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το τριπλό α. Το τριπλό α μας εξασφαλίζει να έχουμε το δυνατότερο χαμηλό κόστος για τη χρηματοδότησή μας. Οπότε αυτό το πολύ χαμηλό κόστος χρηματοδότησης να μπορούμε να το δώσουμε στους πελάτες. Δεν ψάχνουμε να βγάλουμε κάτι από όλο αυτό. θέλουμε οι συναλλαγές να έχουν τέτοια τιμολόγηση που να διασυνδέονται απευθείας με το κίνδυνο. Αν μιλάμε για το εύσιδε και για το υψηλό κινδύνου συναλλαγές, προφανώς δεν μιλάμε για την αδάνεια. μιλάμε για χαμηλή μεν χρηματοδότηση, αλλά θα υπάρχει τέτοια τιμολόγηση που θα είναι ανάλογη με τον κίνδυνο. Και η τιμολόγηση αυτή δεν επιδοτείται. Δεν επιζητούμε λοιπόν το κέρδος, θέλουμε να αναλάβουμε κίνδυνο, οι τράπεζες αναλαμβάνουν κινδύνους και στην ΕΤΕ ακολουθούμε τις επιταγές του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Μέχρι τώρα μας έλεγαν να προσέχουμε τον όγκο, γι' αυτό το είδατε και στην παρουσίαση. Ε, πέρσι δανείσαμε περίπου 80 δις μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας. Είναι τεράστιο ποσό είναι 10 φορέ μεγαλύτερα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Βεβαίω, η Παγκόσμια Τράπεζα ε, λειτουργεί σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, σαφώ. Αλλά αυτό είναι η κανονική μα δραστηριότητα. Και μετά προκύπτει το εξή ερώτημα, ε, ανέκυψε ναι επανειλημμένος. Ποια είναι η διαφορά με το ΕΦΣΥ. Το ΕΦΣΥ έρχεται να συμπληρώσει την συνηθισμένη μα δραστηριότητα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάναμε. Αλλά πέραν αυτού και αυτό είναι το θέμα της προσθετικότητας. Πέραν αυτού και χάρη στην εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο γεγονός και ελπίζουμε ότι η ΕΤΕ θα προβλέψει τα 5 δις για την χρηματοδότηση των δυνατοτήτων του Ταμείου και με αυτά τα 16 συν τα 5 μας θα φτάσουμε στα 21, να μην φτάσουμε να μιλήσω πάλι για τη μόχλευση και τον πολλαπλασιαστή γιατί προκαλεί πολλά ερωτήματα, αλλά να τα δούμε με μία απόσταση. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Δεν είναι ταμείο. Πρώτα απ' όλα, για να τελειώνουμε. Το ταμείο υπάρχει μόνο στο όνομα. Είναι μια διευθέτηση για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΤΕ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, με αυτήν την διευθέτηση, τη συμβασιακή ε, διευθέτηση, ε, ορίζουν ως εγγύηση 16 δις από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 δις για την εξασφάλιση του δυναμικού και μέσω της ΕΤΕ, που είναι ο δικαιούχος της εγγύησης, μέσω της ΕΤΕ λοιπόν, θεωρούμε ότι θα κινητοποιήσουμε 315 δις επενδύσεων την ερχόμενη τριετία από την, ε, στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Είναι πολύ καλό που έχουμε την εγγύηση της Ένωσης, αλλά η ΕΤΕ θα αναλάβει κίνδυνο για την κάθε μια από τις συναλλαγές. Δεν πρόκειται λοιπόν για το ε, αν θα κάνουμε συναλλαγές επειδή έχουμε τις πλάτες της Ένωσης, και δεν θα προσέξουμε όπως παλιότερα την κάθε συναλλαγή μας. Όχι, επειδή ακριβώ έχουμε την εγγύηση της Ένωσης θα μπορέσουμε να καλύψουμε κινδύνους που τώρα δεν μπορούσαμε να τους καλύψουμε Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο της προστατικότητα. Αυτό έρχεται να καλύψει την τακτική μας δραστηριότητα, αλλά μας επιτρέπει κιόλα να καλύψουμε οικονομικές ανάγκες της αγοράς που σήμερα η ΕΤΕ δεν θα μπορούσε να τις καλύψει με το υπάρχον δυναμικό της με τα υπάρχοντα κεφάλαια. Και έτσι φτάνουμε στο πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Επειδή είμαστε τράπεζα και χάρη στην εγγύηση μπορούμε χάρη στο 16 συν 5 21 να κινητοποιήσουμε 60 65 δις στις αγορές κεφαλαίων ε, ή και αξιολόγησης όλος ο κόσμος μας κοιτάει αυτοί που αγοράζουν τα ομόλογά μα ετησίων τέλος πάντων και έχουμε περίπου 80 δι ομολόγων ετησίω και το 30% είναι εκτό Ένωσης, αυτοί όλοι μα εμπιστεύονται διότι θα μπορέσουμε να βασιστούμε σε αυτή την αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση της Ένωσης. Έτσι θα κινητοποιήσουμε 60 δι 60 που θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία. όπω είπε η Μάη, δεν χρηματοδοτούμε ποτέ τα 100% ενός έργου. Το μέγιστο είναι το 50%, το μέσος όρος είναι το 30%, αλλά για το ΕΦΣΥ περιμένουμε να ε, πάμε σε ακόμη μικρότερη συμμετοχή για το καθένα από τα έργα, διότι αυτό που θέλουμε να, μας, να πετύχουμε είναι το επικινδυνότερο τμήμα του έργου. Ε, ο στόχος είναι ακριβώς να συγκεντρώσουμε και γι' αυτό γίνεται το crowding, αυτό χρησιμοποίησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος πάντων κινητοποιούμε θα πει, θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ ρευστότητα εκεί στον έξω κόσμο, στις αγορές. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε έλλειψη ρευστότητας, αυτό δεν ισχύει πλέον. Οι τράπεζες έχουν χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει τέτοια νομισματική πολιτική. Ε, και οι εταιρείε έχουν χρήμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το κρατάνε σφιχτά δεν θα το διαθέσουν στην οικονομία, δεν θα το διαθέσουν για επενδύσεις. Η ε, ΕΤΕ θέλει ακριβώς να βάλει το χέρι στη ρευστότητα που υπάρχει εκεί έξω και στην υλοποίηση των επενδύσεων. Έτσι, λόγω της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι δεν υπήρχε εμπιστοσύνη ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Δεν μπορούμε απλώς να αγαπάμε το παρελθόν, γιατί τότε κρατάμε τις δεκάρες μας και προσιλωνόμαστε σε αυτές και δεν μπορούμε να τις διαθέσουμε. Αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη θέλουμε να δημιουργήσουμε, ότι διαφύγαμε από την οικονομική κρίση, δραπε... Ε, ξεφύγαμε, αλλά θέλουμε να δώσουμε αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα στην οικονομία, για το επίπεδο των επενδύσεων. Τι θέλουμε να πούμε στους επενδυτές. Έχετε εδώ κάποιον στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κιόλα, μιλάμε για την Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε κάποιον που θα αναλάβει ένα μέρος του κινδύνου που έχετε εσείς στις πλάτες σας και θα σας ενθαρρύνει να κάνετε τις επενδύσεις. Μιλάμε για το βασικότερο, το πιο κρίσιμο σημείο του κινδύνου βεβαίω. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλο τον κίνδυνο των επενδυτών. Θα φροντίσουμε λοιπόν να έχουμε συνεργασία μαζί του για να του ανακουφίσουμε αυτόν τον κίνδυνο θα φροντίσουμε οι αγορές κεφαλαίων να συνδυαστούν με τους θεσμικούς επενδυτές και έτσι θα κινητοποιήσουμε το ρευστό. Βλέπουμε ότι ο στόχος είναι να καλυφθούν προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο. Δεν μιλάμε για τα κλασικά δάνεια της ΕΤΕ. Υπάρχει διαφορά λόγω της προσθετικότητας δεν είναι αυτό που σα παρουσίαζε η ΜΑΗ. Αυτό είναι η κανονική μα πολιτική, το τι συμβαίνει συνήθω. Εδώ λέμε ότι με τα ίδια κριτήρια, διότι δεν θα χαλαρώσουμε τα κριτήρια τώρα επειδή κάποιο άλλο αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Ότι τα ίδια κριτήρια αρέσουμε θα υπάρχουν, η ίδια διεξοδικότατη ανάλυση των οικονομικών συνιστοσών, αλλά χάρη στην εγγύηση τη Ένωση θα μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερου κινδύνου. Αυτό που λέμε ουσιαστικά, ε, και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, είναι ότι μπορεί κανείς να διαθετήσει μια ε, συναλλαγή έτσι, ώστε οι πρώτες απώλειες να καλύπτονται από έναν από τους πιστωτές, από ένα κεφάλαιο κινδύνου ή μια εταιρεία. Δεν θα αναλάβουμε αυτές αυτούς τους κινδυνούς, θα πάρουμε ένα πολύ μικρό μέρος, 15-20% και τα υπόλοιπα θα κινητοποιηθούν από την αγορά κεφαλαίων, τους θεσμικούς επενδυτές, με τη ρευστότητα και την διάθεση να λάβουν κίνδυνο. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα του πολλαπλασιαστή, διότι πρώτον θα πάμε από το 21% ε, ως το 60%, από το 21% μάλλον δις το 60%, αλλά αν πετύχει αυτό ε, έχουμε το 20% και το πολλαπλασιάζουμε με 5. Οπότε φτάνουμε στο 315. Αυτό είναι μέσος όρος. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα είμαστε στο 20%. Κάποιες φορές θα αναλάβουμε το 13% και κάποιες φορές 27%. Κάθε φορά αυτό που θέλουμε είναι να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες, ανάγκες του έργου. Θα γίνεται τεχνική και οικονομική ανάλυση, θα κοιτάζουμε το έργο από την πλευρά του περιβάλλοντος, του, του των κοινωνικών οφειλίων, από την πλευρά της οικονομικής ωφέλειας, από την πλευρά του κινδύνου και θα προσαρμόζουμε την παρέμβασή μας στο ελάχιστο. Αυτό που κάνουμε επίτα είναι μετατόπιση στον τρόπο χρήση των δημοσιοκοντιλίων. Οι εγγυήσεις παρέχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το αντιλαμβανόμαστε και είναι πόδινες οι αποφάσεις που λαμβάνονται και αυτό που κάνουμε εμείς είναι για τα έργα που μπορούν να έχουν εμπορική βιωσιμότητα, να γεννήσουν έσοδα δηλαδή για την αποπληρωμή ενός χρέους. Πηγαίνουμε δηλαδή από τις επιδοτήσεις σε κάτι διαφορετικό, διαφορετική χρήση. Θα χρειαστούν κάποια έργα βέβαια μόνο επιδοτήσεις. Και γι' αυτό έχουμε τα διαδρατικά ταμεία και άλλα στοιχεία. Τώρα, πώς γίνεται επιλογή. Όλα τα κριτήρια που ανέφερε η ΜΑΙ θα ισχύουν και για τα έργα του ΕΦΣΙ. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει την ανάλυση. Σας εξήγησε η ΜΑΙ τους τρεις πυλώνες σας είπε πώς αναλύουμε το κάθε έργο με τρεις πυλώνες. Θα δούμε τα οικονομικά αποτελέσματα όχι μόνο του project, αλλά γενικώ πώς θα επηρεάσει την οικονομία εν γέννη και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος και στην κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Θα δούμε τα αποτέλεσματα άμεσα και έμεσα στην απασχόληση, αν προωθεί και πώς προωθεί την επιχειρηματικότητα στην περιοχή και τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, άμεσα, έμεσα, ενεργειακή απόδοση, όλες αυτές τις πτυχές. Θα υπάρχει επενδυτική επιτροπή, Investment Committee. Guarantee Committee, μα, τη λέμε εμείς πιο πολύ, ε, Επιτροπή Εγγύησης. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει ναι ή όχι στη χρήση της εγγύησης αυτή η Επιτροπή. Δεν αποφασίζει ποιες επενδύσεις θα πρέπει ε, ή ποια έργα θα πρέπει να υποστηριχθούν. Αυτό γίνεται από την ΕΤΕ που παίρνει ένα μέρος του ρίσκου όλων αυτών των συναλλαγών και η οποία έχει και όλα τα συστήματα, το προσωπικό, την ε, τεχνογνωσία, την εμπειρία. Εμείς μπορούμε να επιλέξουμε εξαιρετικά, εξαιρετικά άτομα, 6-8 εμπειρογνώμονες εξαιρετικούς που θα πρέπει να γνωρίζουν τους τομείς, αλλά δεν θα μπορούν να κάνουν την ίδια εκτίμηση που μπορούν να κάνουν 300 μηχανικοί. Άρα γιατί να προβούμε σε αλληλεπικαλύψεις αφού τα έχει αυτά η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕ. Άρα την ανάλυση των έργων την κάνει η ΕΤΕ. Κάθε ε, συναλλαγή, κάθε επιχείρηση περνάει από την Επιτροπή Διαχείρισης και το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι κάθε τέτοια δράση είναι μια δράση της ΕΤΕ. Και για να υποφελείται από την εγγύηση θα πρέπει να έχει εγκριθεί όμως και από αυτή την επενδυτική εγκυτική επιτροπή, όπως θέλετε πείτε τη. Θα πρέπει να είναι μια πολύ σαφής απόφαση από την επιτροπή αυτή. Θα πρέπει να πει ναι ή όχι. Δεν μπορεί να πει θα δούμε, θα το αποφασίσουμε ή ας το ξαναδούμε πιο μετά. Γιατί υπάρχει πίσω ένας εργολάβος, ένας ανάδοχος που περιμένει. Αν με επιτρέπετε να μιλήσω εν συντομία για τη σχέση μεταξύ LGTT, εύση και ομολόγων έργων. Υπάρχει η σχέση μεταξύ εύση και LGTT. Περιορισμένα τα ποσά και στενά κριτήρια επιλεξιμότητας. Η διαφορά η μεγάλη με το ΕΦΣΙ είναι ότι εδώ μιλάμε για πολύ ευρύτερα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οπότε έχουμε πρόσβαση σε πολύ διαφορετικά project και μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στις ανάγκες της ε, και, τα προγράμματα στα, ανάγκες της κάθε ε, περιοχής και ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Και με αυτό ολοκληρώνω, εκτό αν υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις που με τα χάρη θα απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πιέζει κάπως ο χρόνος, ε, αν και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και θα χρησιμοποιήσουμε, θα σας χρησιμοποιήσουμε. Θα σας κάνουμε και περισσότερες ερωτήσεις αργότερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε.